Euh, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω να περάσετε καλά στο μεσημεριανό γεύμα και θα ανοίξουμε αυτό τη δεύτερη σύνοδο θέματα απασχόλησης με δύο ουσιαστικά θέματα που έχουν οριστεί και θα σας ε, υπενθυμίσω, είχαμε το αίτημα ενός ε, Γάλλου γερουσιαστή σήμερα το πρωί και άλλα δύο θέματα, συζητήθηκαν με τους ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είχε ξεκινήσει λοιπόν μια διαδικασία για να ακολουθήσουμε, να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα. Το πρώτο φορά την απασχόληση των νέων, το οποίο θα συζητήσουμε μέχρι τις 5 και μετά ένα δεύτερο θέμα, το κοινωνικό αντίκτυπο των προγραμμάτων οικονομικής ε, προσαρμογής στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σε μια εποχή όπου πολλοί συζητούν ε, ε, για τον αντίκτυπο, τον πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας και όπου το διάφορα μέτρα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν τροφοδοτήσει όλο αυτό. Θα συζητήσουμε λοιπόν για να δούμε κατά πόσο όλο αυτό επηρεάζει ή όχι τις πορείες που έχουν χαραχτεί για την κάθε χώρα. Και ειδικότερα θεωρώ ότι ένα από τα διακυβεύματα είναι να επαληθεύσουμε κατά πόσο στο ε, νεαρινή σύνοδο του Συμβουλίου μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πορεία με καθολικό τρόπο, αναγνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτό έχει επιπτώσεις για την ε, κοινωνική κατάσταση, για τις συνθήκες απασχόλησης και για την απασχόληση των νέων. Πριν ξεκινήσουμε αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις ε, γενικού περιεχομένου όσον αφορά τη σημερινή μας συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε, Θέλοντας να βελτιώσουμε τα στοιχεία ενός εξάντε συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, ε, φέτος είναι η τρίτη διαδοχική χρόνια που χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο το οποίο ονομάζουμε Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Το γενικό του πλαίσιο ορίζεται από ένα έγγραφο προσανατολισμού που είναι η αιτήσια επισκόψη της ανάπτυξης. Βάσει αυτής της αιτήσιας επισκόψης της ανάπτυξης, το ΕΡΕΝΟ ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα φέτος 14 Μαρτίου ε, καταλήγει σε γενικούς προσανατολισμούς που στη συνέχεια μεταφράζονται στις ε, ε, απαντήσεις και στις συμβόλες του κάθε κράτους μέλους βάσει αυτών των προσανατολισμών. Αυτό μεταφράζεται σε δύο έγγραφα, το εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που σχετίζονται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλησης που αποτελεί το εργαλείο υλοποίηση του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Το δημοκρατικό ζήτημα φυσικά απαιτεί να επισέρχεται κάθε επίπεδο δημοκρατικής νομιμότητας σε αυτή τη διαδικασία ώστε να δίνει μια άλλη χρειά σε, αυτά, οτιδήποτε, σε όλες τις διαδικασίες της Κομισιόν και σε κάθε διαδικασία που ξεκινά κάθε εθνική κυβέρνηση. Το είχαμε συζητήσει όταν μιλήσαμε για το άρθρο 13 της Δημοσιονομικής Συνθήκης, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Το πώς δηλαδή αυτά τα δύο επίπεδα νομιμότητας κάποια στιγμή πρέπει να συναντηθούν ώστε ο καθένας να ασκεί το δικό του επίπεδο νομιμότητας και δημοκρατικού ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη και την άλλη διάσταση χωρίς απαραίτητα να επηρεάζει την άλλη διάσταση. Τώρα το θέμα που εξετάζουμε σήμερα, την απασχόληση, το κοινωνικό ζήτημα, την καταπολέμηση του αποκλεισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού, αυτό το ζήτημα ε, αντιμετωπίζεται με μεγάλη αποφασιστικότητα. Διότι οι περισσότεροι νόμοι και οι πολιτικοί προσανατολισμοί σε ε, αυτόν τον τομέα εξαρτώνται επίπτωση αρμοδιότητες των κρατών μέλων. Οι οικονομικές πολιτικές έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα επίσης. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ικανότητες όσων ανησυχούν για τα κοινωνικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα στην απασχόληση των πολιτικών που ακολουθούμε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, μας περιέγραψαν σήμερα το πρωί ο Επίτροπος ε, Ρεν και ο Επίτροπος Αντόρ. Τίθε το ζήτημα της ε, ισορροπίας μεταξύ Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Οικονομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου, της ισορροπίας μεταξύ των σχετικών αρμοδιοτήτων και φυσικά σε επίπεδο Συμβουλίου τίθε το ζήτημα ισορροπίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών, το ΕΚΟΦΗΝ, και τη ικανότητα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ που θα συναντηθεί 7 και 8 Φεβρουαρίου για να μιλήσει για την εγγύηση για τους νέους όπου είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένη και όπου θα συμμετέχω αναφέροντάς τους κάποιο κομμάτι των εργασιών μας φυσικά. Η κλασική ανάλυση που οδήγησε στο ερώτημα Μπορεί να ζητήσω σε όσους κάθονται μπροστά είτε να μην μιλάνε, είτε να καθίσουν, είτε να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Το κοινωνικό ζήτημα τίθεται συχνά ως ζήτημα λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ως ε, αποτέλεσμα των αποφασιστικών οικονομικών πολιτικών. Σήμερα παρατηρούμε και θεωρώ ότι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να παρατηρείται το ίδιο που παρατηρούμε και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι όλο και περισσότερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα οποία σχετίζονται με ζητήματα απασχόληση κοινωνικού αποκλεισμού ή ικανότητας ε, ε, αποτελεσματικότητας των κοινωνικών πολιτικών τίθενται ανεξάρτητα από τους οικονομικούς προσανατολισμούς που τίθενται. Το απλό σλόγγαν ότι όσο περισσότερες επενδύσεις έχουμε και όσο περισσότερες αναπτυξιακές πολιτικές τόσο το καλύτερο δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής όπως αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Και αυτό είναι ένα από τα διακυβεύματα των δύο θεμάτων που έχουμε να μελετήσουμε σήμερα μαζί, σήμερα το απόγευμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με την κατάσταση της απασχόλησης και σε σχέση με την ενέργεια των νέων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζετε τα σχετικά νούμερα και δεν θέλω να μακρηγορήσω με τέτοια στοιχεία. Πολύ απλά θα ήθελα να σας πω ότι κατά την πρώτη μας στρογγυλή τράπεζα που θα αφορά το ζήτημα της απασχόλησης των νέων και που θα ξεκινήσουμε αμέσως. Θα μιλήσουν δύο πρόεδροι επιτροπών. Ο Έλληνας ε, πρόεδρος ε, που είχαμε την τύχη να συναντήσουμε ορισμένοι από μας χθε, ο κύριος Κρεμαστινός. Και μετά για εκ μέρους της Ισπανίας, ε, ο κύριος Άσπυρος Βλάρ, Σας, σας εύχομαι, σας καλωσορίζω σε ευθύνη μα εδώ τη συνεδρία και μετά όσον αφορά την εγγύηση για του νέου, έτσι όπω υλοποιείται σε μία από τι χώρε που πάντα δίνονται ω υπόδειγμα, έχουμε την τιμή και την ευχαρίστηση να έχουμε εδώ την πρόεδρο τη Επιτροπή Απασχόληση ε, του Φιλανδικού Κοινοβουλίου, κ. Φιλανδόφ, και θα σα δώσω το λόγο στο τέλο αυτών των παρουσιάσεων και θα ολοκληρώσουμε με του δύο εισηγητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου ευχαριστώ για την παρουσία του από την αρχή των εργασιών μας, την κυρία Στρίσλευσκα και τον κύριο Κρίστινσεν. Η, η κυρία πρόκειται από το Έλκο και ο κύριο Κρίστινσεν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ώστε να έχουμε ισορροπία. Δυο λόγια πριν σας δώσω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Φυσικά για να σας υπενθυμίσω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Αντόρ με την υποστήριξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετήσαμε ένα κείμενο το οποίο θα βρείτε στους φακέλους σας με το οποίο ζητάμε το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ που θα συναντηθεί 7 και 8 Φεβρουαρίου να λάβει υπόψη πλήρω τι προτάσει αυτέ για την εγγύηση για του νέου. Τι είναι η εγγύηση για του νέου, Είναι η ιδέα ότι ένα νέο, ο οποίο χάνει τη δουλειά του, ο οποίο ε, ε, έχει μόλι πάρει πτυχίο, έχει μόλι ολοκληρώσει την κατάρτιση, δεν μπορεί να παραμείνει πάνω από τέσσερι μήνε σε μια άνεργο, χωρί να του προταθεί μία λύση αντικατάσταση κάποια άλλη κατάρτιση, κάποια δουλειά, κάποιο είδου μαθητεία. Η πρόταση έτσι όπω την υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε μία χρηματοδότηση βάσει των αναγκών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό προποθέτει ότι εφόσον τα κράτη-μέλη αποδεχθούν την πρόταση της Κομισιόν ώστε να οριστεί η συμμετοχή του ως 25% στην πολιτική συνοχής. Πρέπει να σας πω όμως ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκεφτήκαμε ότι το ιδανικό και το ιδανικό σου μπορεί να επιτευχθεί αμέσως το ιδανικό θα ήταν αυτή η εγγύηση για τους νέους να χρηματοδοτείται από ένα ειδικό δημοσιονομικό κονδύλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο κατά κάποιον τρόπο θα έχει ως αποτέλεσμα ότι η εγγύηση για τους νέους ε, δεν θα αποτελεί απλά το, ένα ελάχιστο δικαίωμα αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πέραν και αυτής της κοινωνικής αναγνώρισης θα αποτελούσε ένα εργαλείο καθοδήγησης και συμβολής ενό τέτοιου παράγοντα, ο οποίο θα θεωρηθεί αυτόματο σταθεροποιητικό παράγοντα ουσιαστικά και θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο συνένεση αυτή η μορφή αποζημίωσης ας πούμε. Ε, έπρεπε λοιπόν να τα πω όλα αυτά, φυσικά μακρηγόρησα. Δεν σας παροτρύνω να ακολουθήσετε το παράδειγμα μου, σας δίνω αμέσω, κύριε Κρεμαστίνε το λόγο για να μας μιλήσετε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο στη δική σας χώρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα μέτρα για την απασχόληση των νέων και επίσης να μας μιλήσετε για τις προοπτικές που βλέπετε όσον αφορά αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική για μια εγγύηση για τους νέους. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Oh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Όπως και χθε θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Όπως γνωρίζετε, η παγκόσμια οικονομική κρίση ε, εκφράζεται σήμερα σαν οικονομική ευρωπαϊκή κρίση και αντικατοπτρίζεται ε, καλύτερα στις χώρες του Νότου με κατεξοχήν, κατεξοχήν την Ελλάδα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί τελικά σε πολλά κακά ανεπιθύμητα αλλά ένα από τα χειρότερα είναι η ενεργεία και ειδικότερα η ενεργεία των νέων που αν δει κάποιος και μελετήσει τα στοιχεία της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα ε, θα καταλάβει τι περίπου συμβαίνει στο διεθνώς γίγνεστη. Ε, σήμερα η Ευρώπη έχει πάνω από 25 εκατομμύρια ανέργους. Ε, η Ελλάδα έχει πάνω από το 30% του πληθυσμού της με επίσημα στοιχεία που τον φέρνουν γύρω στο 25 με 26%. Και το νέο η ανεργία στην Ελλάδα με επίσημα στοιχεία ξεπερνάει το 50%. Ε, το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της ανεργίας. Δηλαδή από τρίμηνο σε τρίμηνο η ανεργία αυξάνεται δραματικά και δεν δείχνει ακόμα τάση ε, εξισορρόπησης. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το τρίτο τρίμηνο του 12 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.739.000 και των ανέργων σε 1.123.000. Το ποσοστό της ανεργίας το τρίμηνο από 24,8 από 23,6 ανήλθε στο 24,8 μέσα σε ένα τρίμηνο. Και αυτό είναι, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 8,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ρυθμός της ανεργίας καλπάζει. Αποτέλεσμα, τελικό αποτέλεσμα είναι η ανεργία αλλά στην ενεργεία οδήγησαν μέσα στα δύο τελευταία χρόνια δύο σημαντικά γεγονότα. Η απότομη, θα έλεγα, η δημοσιονομική, η αυστηρή ε, δημοσιονομική πολιτική χωρίς ανάπτυξη και υψηλή φορολογία. Αυτό οδήγησε σε μια πρωτοφανή ύφεση με λάτωση του ΑΕΠ κατά 4 έως 6% με αποτέλεσμα να κλείσουν οι επιχειρήσεις μαζικά και η χώρα να οδηγηθεί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα σε μια κατάσταση φτωχοποίησης. Εκείνο δε το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό και αν θέλετε ε, δεν υπήρχε, υπήρξε προστασία από μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλα τα πέριξ της Ελλάδας ε, κράτη ε, είχαν, έχουν ένα ΑΕΠ πολύ χαμηλό έχουν πολύ χαμηλή φορολογία με αποτέλεσμα μαζικά όλες οι επιχειρήσεις που είχαν έδρα τους στην Ελλάδα να μετακομίσουν στις διπλανές χώρες. Αποτέλεσμα ε, ουσιαστικά να κλείσει η μία μετά την άλλη σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτής της ανεργίας είναι ότι το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών είναι σημαντικά ψηλότερο σε σχέση με τον ανδρών. 28 προς 21. Και το υψηλότερο ποσοστό της ανεργίας, όπως είπαμε, 56,6% παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών. Εκείνο που είναι επίσης ενδιαφέρον και πιθανόν να αντιμετωπίζεται και στις άλλες χώρες είναι ότι η, το μεγαλύτερο ποσοστό της ανεργίας αφορά εκείνους που δεν διαθέτουν γνώσεις βασικής παιδείας. Αντίθετα, αυτοί που έχουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης έχουν ποσοστό ανεργίας 28% ενώ αυτοί που δεν έχουν καθόλου βασική εκπαίδευση η ανεργία τους ανέρχεται στο 41%. Ενώ αντίθετα επίσης στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ποσοστό της ανεργίας υποχωρεί στο 12,6 περίπου το ποσοστό των νέων ανέργων, δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην εργασία, ανέρχεται σε 24,7% του συνόλου των ανέργων. Ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί δηλαδή που αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες, αποτελούν το ανησυχητικό 52,6%. Αντίστοιχα στην Ευρώπη, 11 εκατομμύρια άνεργοι ε, είναι άνεργοι εδώ και ένα χρόνο. Εκείνο που είναι επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι σε περιοχές που υπάρχουν υποδομές έχουμε χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους που σε ποσοστά που κυμαίνονται από 11 έως 13%. Και το χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο ότι υπάρχουν υποδομές, υπάρχει τουρισμός και απασχολούνται ο πληθυσμός. Ενώ αντίθετα στις άλλες περιοχές της χώρας το, πληθυ... ποσοστό της ανεργίας καλπάζει πολύ πάνω από το μέσον όρο. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη των υποδομών και στις περιοχές ακόμα αυτές όπως είναι οι μαρίνες, η αξιοποίηση των ακτών στα μικρά νησιά αλλά και στις βιομηχανικές χώρες ε, που έχουν βιομηχανικά προϊόντα για εξαγωγή. Ε, η ανάπτυξη των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε καλύτερες μέρες από πλευράς ανεργίας ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ελληνικής ανεργίας, η Ελλάδα σήμερα εφαρμόζει σταδιακά μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης με τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας στις 10 του Ιανουαρίου αυτού του μήνα ε, που θέλει προγράμματα δράσης και απασχόλησης των νέων τα οποία συμβαδίζουν ε, με τα, με, τα αποτελέσματα τα ευρωπαϊκά. Η εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι υποδομές αποτελούν βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της, της ανεργίας και συμπερασματικά θα έλεγα ότι η ανάδειξη της αναγκαιότητας αυτής να υποστηριχθούν οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με τη σταδιακή εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της νεανικής απασχόλησης θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου για την κλιμακούμενη αλλά σταθερή καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ. Euh. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρεμαστινέ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. <clears throat> Πρωτού δώσω το λόγο τώρα στον ε, συνάδελφο τον κύριο Ασπυρός Φιγιάρα από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει ένα φύλλο χαρτί στο οποίο μπορείτε να εγγράψετε το όνομά σας, εάν θέλετε να λάβετε το λόγο, στο, για το πρώτο θέμα ή για το δεύτερο θέμα του απογεύματος και για τα δύο. Και έχετε επίσης και μία σύντομη σύνοψη των εννέα συμβολών που έχουμε λάβει από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τα θέματα αυτά, τις τρεις φορές, και τα κείμενα <clears throat> βάσης, κείμενα αναφοράς, που είναι τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχει και η έκθεση της κυρίας Λοπές Φοντανιέ που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό έγγραφο και αντιμετωπίζει τα θέματα απασχόλησης και ανάπτυξης. Με έναν τρόπο ίσως διαφορετικό από ό,τι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο μιλητή μας και δίνω μέσα στο λόγο στον κύριο Χωσέ Εουχένιο Ασπυρός Φιγιάρ από την Επιτροπή, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία αυτή που μου έδωσε να συμμετάσχω στην σημερινή συνεδρίαση. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ καλό βήμα για τη συζήτηση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα της ανεργίας των νέων είναι πάρα πολύ οξύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ένα θέμα που έχει δραματικές διαστάσεις σε χώρε όπως η Ισπανία, η δική μου χώρα, όπου η ανεργία των νέων μεταξύ 16 και 30 ετών ξεπερνάει το 55%, ενώ είναι μόνο 25% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε δηλαδή για 7,5 εκατομμύρια νέων από 16 έως 25 ετών που δεν είναι ούτε σε κάποιες σπουδέ ούτε εργάζονται. <clears throat> Στι 5 Δεκεμβρίου του 2012 η Κομισιόν ενέκρινε μια πρόταση σύσταση προ το Συμβούλιο για τη δημιουργία της λεγόμενης εγγύησης των νέων, στην οποία αναφέρθηκε και η πρόεδρό μας, και η οποία έχει υποστηριχθεί από το Εβραίο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τη 16η Ιανουαρίου 2013. Ποια είναι τώρα η θέση τη Ισπανία σε σχέση με την απασχόληση και την εγγύηση για του νέου. Καταρχήν, μέσα στα πλαίσια τη ε, συνολική πολιτική προσέγγιση και τη μακροοικονομία, είναι σημαντικό το πακέτο μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Ραχώη από το Παρτίδο Ποπουλά για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος, για την λιτότητα και τη διαφάνεια του προϋπολογισμού, την συμπίεση των δαπανών, τη μεταρρύθμιση του τραπεζο, πιστοτικού τραπεζικού τομέα, του αγώνα κατά των ε, πτωχεύσεων, του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και, της, ε, ε, και των παροχών που δεν έχουν δικαίωμα δικαιούχοι σε αυτές, τη μεταρρύθμιση της παιδεία, την ενότητα της αγοράς και επίσης την ε, μείωση των ε, αποδοχών των υπαλλήλων της κυβέρνηση. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν στη σταδιακή υπέρβαση της κρίσης και στην εκ νέου δημιουργία πλούτου και απασχόλησης και για τους νέους. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και ένα δεύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων στον εργασιακό τομέα. Η μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό είχε σαν γενικό χαρακτήρα να υπάρξει η χρήση της ευκαμψίας η οποία θα πρέπει να αντικαταστήσει μια απλή και μόνο καταστροφή θέσεων εργασίας. Το 2012 υπήρξαν μέτρα για να μπορέσει να διατηρηθεί η απασχόληση σε, σε καιρό κρίσης με μείωση των αποδοχών και της εργασιακής ημέρας και εβδομάδος, μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη κατάρτιση, παραγωγικότητα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. Και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια καλύτερη πρόταση παρά η απλή απόλυση. Υπάρχουν διάφορα σημαντικά ε, σημαντικοί εργοδότες όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν συμμετάσχει σε αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν υπάρχει το συμβόλαιο των, το λεγόμενο συμβόλαιο των εργοδοτών είτε είναι ε, απεριορίστου χρόνου, είτε όχι. Σε 10 μήνες μέσα έχουν υπάρξει 35.000 περίπου τέτοια συμβόλαια για νέους κάτω των 30 ε, ετών, περίπου 45%. Και επίσης έχουν εγκριθεί ε, 150 προγράμματα το 2012 και 59 το 2011. Επίσης, με το βασιλικό διάταγμα της 8ης Νοεμβρίου θεσπίζεται το, το συμβόλαιο για την κατάρτιση και τη μαθητεία και το διάταγμα αυτό καθορίζει τις βασικές αρχές αυτού του προγράμματος. Από το Μάρτιο στο Δεκέμβριο του 2012 το, τα συμβόλαια αυτά ε, μαθητείας και κατάρτισης έχουν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με το 2011 και έχουν φτάσει στα 6.584 συμβόλαια αυτού του είδους, συμβάσεις αυτού του είδους καλύτερα και ουσιαστικά διπλασιάστηκαν τα συμβόλαια για τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο κατάρτιση που πέρασαν από 6.182 σε 13.259. Ξέρω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνουν και τα θέματα μείωσης της ανεργίας των νέων <clears throat> και οδήγησαν σε 30.000 δημιουργίες θέσεις απασχόλησης για νέους κάτω των 25 ετών, αυτά φαίνονται ίσως περιορισμένα μέσα στο πλαίσιο της μαζικής ανεργίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά δείχνουν και μια αλλαγή στην τάση που παρουσιάζεται και μια πρώτη, ένα πρώτο ψήγμα ελπίδας για το μέλλον. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Το, σχέδιο απασχόλησης του 2012 έχει ένα από τους έξι στόχους του, την μείωση της ανεργίας των νέων και θεωρεί ότι με μια σειρά από μέτρα τα οποία παρέχουν ε, κίνητρα για την καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση για τις ε, καλύτερες πρακτικές επιχειρήσεις στις, ε, στα κίνητρα για μια ε, αορίστου χρόνου σύμβαση εργασία και την εργασία των νέων, όλα αυτά θα βοηθήσουν την κατάσταση. Έχουμε στο τρίτο σημείο, την δονή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι υποδιαπραγμάτευση στους κοινωνικού εταίρους η στρατηγική ε, εργοδοσία και απασχόληση των νέων και περιλαμβάνονται όχι μονάχα δράση τη δημόσια αρχή, αλλά και των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων και φυσικά και του ιδιωτικού τομέα. Με αυτέ τι ε, ενέργειες μπορούν να συμμετάσχουν, σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που θέλουμε. Η στρατηγική αυτή έχει σαν στόχο να ενισχύσει την εγγύηση για τους νέους και να ενισχύσει τα υπόλοιπα στοιχεία αυτή τη σύσταση, κυρίω για να εξασφαλιστούν ότι όλοι οι νέοι μέχρι 25 ετών θα έχουν μια προσφορά εργασία ποιότητα ή κατάρτιση ή επιμόρφωση, μαθητεία ή πρακτική εξάσκηση μέσα στου τέσσερι μήνε που ακολουθούν την ανεργία του ή το τέλο τη ε, εκπαίδευσή του. Όπω ελέγχθηκε σήμερα το πρωί, στη Μαδρίτη είχε γίνει μια συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Συνδικάτων πρόσφατα, όπου η, η Φάτιμα Μπάνιας, η υπουργό Απασχόλησης της ε, ε, Ισπανίας, ανακοίνωσε μια μείωση των κοινωνικών εισφορών για τους ε, εργαζόμενους και επίσης 30% μείωση της φορολογίας τους για τους νέους κάτω των 30 ετών στους πρώτους 24 μήνες της απασχόλησής τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να γίνει δυνατό να αντιμετωπιστεί η ανεργία ως και μια ευκαιρία για αυτοαπασχόληση και θα υπάρξει και η δυνατότητα για νέες οικονομικές δράσεις στον τομέα αυτό. Τέλος, μπορώ να θέσω και μια προσωπική νότα, τα δικά μου συμπεράσματα. Παρά το γεγονό ότι η σύσταση τη Κομισιόν αντιμετωπίζει θέματα όπω το θέμα του αποκλεισμού των νέων από το χώρο εργασία, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο τη λεγόμενη χαμένη γενιά. Με ιδιαίτερα μέτρα υπέρ αυτών των νέων και ακόμα των λιγότερων νέων. Πολλοί από του οποίου είναι άνεργοι μακρά διαρκεία και δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να είναι πράγματι μέσα στην αγορά εργασία και επομένω πλήττονται και από τι ψυχολογικέ συνέπειε είναι η άλλη όψη του συνδρόμου απανθράκωσης ή burnout, αυτών οι οποίοι έχουν εργαστεί πάρα πολύ. Είναι αυτοί που δεν έχουν εργαστεί καθόλου και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και ο κύριος Επίτροπος Απασχόλησης ανέφερε το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θεωρώ λοιπόν εν κατακλείδη πάρα πολύ σημαντική την σύσταση την οποία συζητούμε. Είναι μια απάντηση που την περιμένουν με αδημονία οι νέοι μας και είναι απαραίτητη για την κοινωνία μας και με μέτρα αυτού του είδους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κάποια απάντηση στην τραγωδία και τη μάστιγα αυτή που έχουν να αντιμετωπίζουν οι νέοι με την ανεργία. Θα πρέπει να συναρμοστεί φυσικά και με πολιτικέ οικονομική ανάπτυξη, όπω έχουν πει πολλοί ευρωβουλευτέ και εθνικοί βουλευτέ, ώστε τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να καταφέρουν την υπέρβαση αυτή τη κρίση. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφε, για όλες αυτές τις διαφωτιστικές πληροφορίες. Δίνω τώρα το λόγο στη συνάδελφα μας κυρία Φιλατόφ, Πρόεδρο της ε, Επιτροπής Απασχόλησης και Ισότητας του Φιλανδικού Κοινοβουλίου, όπου εγγύηση για τους νέους έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του benchmark ε, ή της εκμάθησης μέσω της πράξης. Ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε για την εμπειρία σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα γνωρίζουμε όλοι ότι για, την, για το μέλλον της κοινωνίας η απασχόληση των νέων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένας άνεργος νέος κοστίζει στην κοινωνία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Η ε, κυρία Φιλάτοφ παρακαλείται να βγάλει τα ακουστικά της, γιατί υπάρχει αντίχηση. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Και κα... okay. Pyrin puhumaan siitä suhteellisen konkreettisesti, koska luulen, että sitä kautta puheenvuorostani on eniten. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται. Καταρχάς, ο πρώτος πυλώνας της πολιτικής μας είναι ο εξής. Οι νέοι μέχρι 25 ετών ή οι απόφοιτοι μέχρι 30 ετών πηγαίνουν στα κέντρα βρέσεως εργασίας και προσπαθούν αυτά να τους βρουν ε, δουλειά όσο το δυνατόν συντομότερα. Έπειτα τα κέντρα αυτά διασφαλίζουν την ε, κατάρτιση για όλους ε, όσους έχουν βασική εκπαίδευση. Αυτό ήταν ο δεύτερο πυλώνας. Και ο τρίτο πυλώνας είναι ή εξαφανισμένοι όπως τους λέμε. Είναι νέοι άνθρωποι που δεν ε, έχουν κάποια κατάρτιση, που δεν αναζητούν εργασία στα γραφεία βρέσος εργασία. Ορισμένοι από αυτούς ε, προσέχουν μικρά παιδιά στο σπίτι, όμως πολλοί βρίσκονται σε συνεχιζόμενη απειλή κοινωνικού αποκλεισμού. έχουμε αναλάβει δράσεις έτσι ώστε να τους εντάξουμε πάλι στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Είμαστε πολύ κοντά στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη. Το σκεπτικό είναι για ένα σχέδιο απασχόλησης το οποίο θα συντάσσεται για κάποιον άνεργο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που εκείνος αναζητεί εργασία επίσημα. Και μέσα σε τρεις μήνες ο νέος αυτός είτε έπρεπε να έχει λάβει κάποια μορφή απασχόλησης, πληρωμένης εργασίας, είτε μαθητείας, είτε κάποια άλλη μορφή ε, δραστηριότητας, έτσι ώστε να αποτραπεί ο αποκλεισμός του και να σταματήσει να είναι άνεργος. Πέντε μήνες ανεργίας είναι ένα πολύ σοβαρό χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα κινδυνεύει ο άνεργος από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε την, ε, το πρόγραμμα εγγύηση για τους νέους έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όσο δυνατόν περισσότεροι νέοι στην αγορά εργασίας. Έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται κάρτα Σάντσι», το οποίο χρησιμοποιούν οι νέοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασία, για να βρουν δουλειά σε μια εταιρεία. Ε, το πρόγραμμα αυτό έχει ως εξή. Η εταιρεία για να προσλάβει τον άνεργο μπορεί για διάστημα μέχρι 10 μήνες να λαμβάνει επιχορήγηση από το κράτος ύψους μέχρι 700 ευρώ. Αυτό είναι μια ευκαιρία για τους νέους και να μπουν στο κλίμα της θέσης εργασίας, αλλά και για την ίδια την εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί μετά να προσλάβει τον νέο υπό διαφορετικές συνθήκες με πλήρη απασχόληση. Επίσης, όσον αφορά τους απόφοιτους, που είναι πάνω από 25 ετών και δεν μπορούν να βρουν εργασία, τους παρέχεται ειδική υποστήριξη έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Το σκεπτικό πίσω από αυτό το πρόγραμμα είναι να γίνουν περισσότερο αποδοτικές οι υπηρεσίες ε, προς τους νέους αυτούς και αυτοίωση ανάμεσα στους οργανισμούς που βοηθούν τους νέους να βρουν δουλειά και να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη κατάρτισης από την οποία υποφέρουν πολλοί νέοι. Όποιος νέος έχει συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε κατάρτιση. Και διευκολύνεται η πρόσβαση ιδιαίτερα σε εκείνους που δυσκολεύονται να βρουν κάποια θέση επαγγελματικής ε, κατάρτισης. Ιδιαίτερα οι νέοι ενήλικες οι οποίοι έχουν εισέλθει μεν στην αγορά εργασίας, δεν έχουν όμως κάποια μόνιμη απασχόληση. Για τους νέους αυτούς προσπαθούμε να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να βρουν αυτήν τη δουλειά, αυτήν την πλήρη απασχόληση. Και η επαγγελματική κατάρτιση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όσο περισσότερη κατάρτιση και υψηλότερη εκπαίδευση διαθέτει κάποιος, τόσο καλύτερες είναι και οι πιθανότητες του να βρει δουλειά. Έχουμε δει ότι αυτοί που επωφελήθηκαν περισσότερο από το πρόγραμμα αυτό είναι οι νέοι που βρίσκονται πολύ κοντά στην αγορά εργασία, που έχουν καλέ δεξιότητε και αυτό που κάναμε εμεί είναι να είμαστε περισσότερο προορατικοί και να έχουμε περισσότερο θετική αντιμετώπιση στα μέτρα που υιοθετούμε. Ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ε, προβλήματα εξάρτησης, από ουσίες, διανοητικής υστέρησης. Ή νέοι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει το σχολείο πολλές φορές. Για παράδειγμα, εάν κάποιος νέος δεν πάει στο σχολείο μία μέρα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα πάει στο σπίτι, θα του χτυπήσει την πόρτα και θα φροντίσει ώστε να επιστρέψει στο σχολείο, έτσι ώστε ο νέος αυτός να τελειώσει το σχολείο και να έχει πιθανότητες μετά να βρει δουλειά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της ε, δικτύωσης και της σύνδεσης ανάμεσα στις κοινωνικές ε, υπηρεσίες πρόνοια και στις υπηρεσίες απασχόλησης και στις άλλες τοπικές αρχές. Σημαντικό στοιχείο αυτών των μέτρων είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Οι προθεσμίες δεν είναι τόσο σημαντικές όσο η συνεχής παρακολούθηση και η παρακολούθηση κατά περίπτωση, ανάλογα τον άνθρωπο. Και είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τη γενική εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ε, μας δώσετε πολύ ακριβείς πληροφορίες και πολύ λεπτομερείς. Θα ήθελα να καταχρηστώ του προνομίου μας Προέδρου για να σα κάνω μια ερώτηση. Σε ποιο δημοσιονομικό κονδύλιο, με ποιο μάλλον κονδύλιο χρηματοδοτούνται τα 700, καταβάλλονται τα 700 ευρώ ω συμπλήρωμα για τη ε, μη δυνατότητα καταβολή ε, επαρκών μισθών από ορισμένε επιχειρήσεις όπως προβλέπετε από τις λογικές συμβάσεις. Σε ποιο κονδύλιο λοιπόν εντάσσονται αυτά τα 700 ευρώ, από ποιο χρηματοδοτούνται. Πολύ καλή ερώτηση. Το Υπουργείο Εργασία έχει ένα κονδύλιο του προϋπολογισμού για εκπαίδευση ανέργων, υποστήριξη προς άνεργους. Αυτά τα χρήματα προέρχονται από αυτή την ίδια γραμμή του προπολογισμού. Αυτό αποφασίζεται από το κέντρο εργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω τώρα το φοβερό καθήκον κατανομής του δικαιωμάτους ομιλίας. Πριν δώσω το λόγο, μάλλον θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας δώσω το λόγο μετά. Δίνω πρώτα λοιπόν το λόγο στην κυρία Σδρίσλευσκα, κυρία εισηγήτρια για το θέμα της απασχόλησης των νέων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή τη συνάντηση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που αφιερώνουμε χρόνο σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ άλλων στους νέους στην αγορά εργασίας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι οι λύσεις που υιοθετούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι απλά συστάσεις. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που πρέπει να δρουν και να εφαρμόζουν πρακτικά αυτές τις ιδέες, καθώς και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που εδώ βρίσκονται βουλευτές από τα κράτη-μέλη. Η κατάσταση για τους νέους αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα εξαιρετικά δύσκολη. Η οικονομική κρίση την οποία εφίσταται η Ευρώπη έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμφάνιση νέων θέσεων εργασίας. Οι εργοδότες προσπαθούν να μειώσουν το κόστος των εργατικών Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, το 40% των ανθρώπων με βραχυ... βραχυπρόθεσμες συμβάσεις είναι νέοι. Δεν είναι πολύ αισιόδοξη η κατάσταση όταν νέοι άνθρωποι... Δεν είναι μια πολύ καλή προοπτική για ένα νέο. Δεν πρέπει επομένως να ξεχάσουμε και το σημείο αυτό και φυσικά και η δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη έχει συμβάλει στο ότι για τους νέους να είναι όλο και πιο δύσκολο να μπορούν να έχουν μια οικογένεια. Γιατί αυτοί οι νέοι δεν έχουν καμιά προοπτική για επαγγελματική αποκατάσταση και επομένως είναι υποχρεωμένοι να αναβάλουν πάντα την απόφαση για τη δημιουργία α, Έχουν γίνει τώρα όλες αυτές οι ενέργειες το πακέτο για την απασχόληση των νέων, για την ε, κατάρτιση των νέων και επίσης το πακέτο, η πρόταση αυτή για την εγγύηση των νέων. Αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως όλα αυτά τα στοιχεία. Τα αποτελέσματα δεν έχουν εξάλλου αποδειχθεί ιδιαίτερα θετικά. Γι' αυτό <clears throat> νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο σε μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη αυτά τα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αποδίδουν καρπούς αυτά τα μέτρα. Και αυτό το θέμα διαλαμβάνω στην έκθεσή μου για τους νέους στην αγορά εργασίας. Έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι στην ανάλυση της κατάστασης των νέων δεν πρέπει να λησμονήσουμε το γενικό οικονομικό πλαίσιο και την γενική ανεργία η οποία σοβεί στην Ευρώπη. το ποσοστό των ανέργων έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά επίσης αυξάνει και το, ο αριθμός αυτών οι οποίοι ενώ έχουν μακρά προϋπηρεσία και πείρα απολύονται. Αυτοί δεν μπορούν να ανοίξουν θέσεις για τους νέους γιατί οι θέσεις τους δεν μπορούν να καλυφθούν από νέους. Δεν δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης επομένως για τους νέους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υποστηριχθούν από, δημόσιο, από το δημόσιο τομέα, από τις κυβερνήσεις, μέτρα τα οποία προωθούν άμεσα τις ε, θέσεις απασχόλησης των νέων. Η δε διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν ήδη θα πρέπει να εξασφαλιστεί με κίνητρα προς τους ε, εργοδότες, οι οποίοι ήδη οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν τα κίνητρα για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η εγγύηση αυτή για τους νέους, για μαθητεία, για επιμόρφωση, για κατάρτιση, και τα λοιπά για τους νέους που είναι μέχρι 25 ετών και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 30 ετών. Αυτή η εγγύηση των νέων είναι μια σημαντική πολιτική όθηση η οποία μπορεί να δοθεί. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων απασχόλησης και των φορέων κατάρτισης και επίσης και η συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις των νέων που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά. Εγώ θεωρώ θετικό ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ακολουθήσει και ορισμένες κατευθύνσεις και προτάσει που δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση τη Κομισιόν και έχουν ενισχύσει τι δυνατότητε τοπική απασχόληση. Συγχρόνω όμω θα ήθελα να κάνω και μία έκκληση προ τα κράτη-μέλη να μην παραμείνουν αδρανοί χρησιμοποιώντα ω πρόσχημα την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και έτσι να παραγνωρίσουν την ανάγκη υποστήριξης μέτρων για την ε, απασχόληση των νέων. Έχουμε όλη αυτή τη γενιά λοιπόν νέων που δεν είναι σε κάποια εργασία, σε κάποια κατάρτιση ή σε κάποια μαθητεία. Μιλάμε για ένα των 15% μάλλον των νέων στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους νέους οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν δυσκολία να αντιμετωπίσουν το χώρο εργασίας. Είναι απαραίτητο για αυτό το λόγο να εξυγχρονίσουμε το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει ένα <clears throat> μοχλό για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Θα πρέπει επίσης και η εκπαίδευση και η κατάρτιση να αντιμετωπίσουμε περισσότερο τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι εργοδότες θα πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο για την προσέλκυση ταλαντούχων νέων και οι νέοι θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να ξέρουν με ποιο τρόπο θα μπορούν να βρουν εργασία σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή επίσης πώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρχουν και προτιμησιακές ε, δυνατότητες για τους νέους παραδείγματο χάρη με φορολογικά κίνητρα για να προχωρήσουν σε μια τέτοια δημιουργία επιχείρηση. Στην Πολωνία έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και έχουμε προχωρήσει στην ε, εκπόνηση μιας μεταρρύθμισης στον εργασιακό τομέα. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται για να βοηθήσουν την, το σχεδιασμό της καριέρας των νέων και ο στόχος μας επίσης είναι να δώσουμε κίνητρα με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και να έχουμε και μεγαλύτερο έργο στην αγορά εργασίας. Και όταν πρόκειται για, τις, ε, για την πρακτική εξάσκηση των νέων, στην Πολωνία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμβάσεις με τους νέους, το οποίο βέβαια δεν επαρκεί για να εξασφαλίσουν όλοι αυτοί οι νέοι μία θέση εργασίας. Επομένως είναι πάρα πολλά τα οποία εξαρτώνται από την υποστήριξη που δίνει το κάθε κράτος μέλος, αλλά συγχρόνως και από την ε, ικανότητα του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε τελική ανάλυση και από την προσωπική πρωτοβουλία των νέων οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν μια, ένα, μια επαγγελματική κατεύθυνση. Έχουμε ένα... Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή στην Πολωνία και είναι το 23% του τον ε, ναι, στην Πολωνία. Η κατάσταση δυστυχώς είναι ακόμα τραγικότερη. 28% ε, των νέων είναι άνεργοι. Και αυτοί οι νέοι δεν έχουν καμία δυνατότητα ούτε να βρουν ε, δουλειά και πολλές φορές απογοητεύονται, εξοργίζονται και εγκαταλείπουν τις προσπάθειες. Πιστεύω πως πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε δράση έτσι ώστε να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφο. Την τελευταία εισαγωγική ομίλια θα δώσει ο συνάδελφος κύριος Κρίστενσεν για την στρατηγική για την νεολαία 2012. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα επί αυτού του εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος της ενέργειας των νέων. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους νέους της. Έτσι έγραψε η Επιτροπή στην εκθεσή της του 2009 και πιστεύω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα διαμορφωθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στους νέους να συμβάλλουν στο μέλλον της Ευρώπης. 22,8 των νέων της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, δηλαδή 5,5 εκατομμύρια νέοι. Και μάλιστα πολλοί νέοι αισθάνονται ότι κάποιος τους στερεί το μέλλον τους. Πολλές προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Τις οικονομικές προκλήσεις, την οικονομική κρίση, την ανταγωνισμό από τις άλλες χώρες. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται κάτι να διορθωθεί στα γρήγορα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική στρατηγική για τους νέους. Ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η προσέγγιση μας προς τους νέους θα είναι συντεταγμένη. Θα χρειαστούμε συντονισμένες προσπάθειες η στρατηγική για τους νέους ε, της Κομισιόν από το 2010 έως το 2018 είναι μια άριστη στρατηγική. Βρισκόμαστε στο πέρας της πρώτης τριετίας και είναι κατάλληλη στιγμή για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι όπως φαίνεται η στρατηγική αυτή έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει εθνικές στρατηγικές για τους νέους που εστιάζονται στην κοινωνική ένταξη των νέων και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού. Είμαι ιδιαίτερα επίση ικανοποιημένο με το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ακροάσει με του νέου σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο ενό διαρθρωμένου διαλόγου. Δεν σε ολόκληρη την Ευρώπη φυσικά. Οι νέοι είναι εκείνοι ενδιαφερόμενοι του όλου ζητήματο. Κοιτώντα λοιπόν αυτόν τον τριετή κύκλο που έχει μόλις κλείσει, πρέπει να αξιολογήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, σε ποιους τομείς θα εστιαστούμε στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Επίσης, σε αυτή τη χρονική στιγμή θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα δεν ήταν επαρκή για την αντιμετώπιση της γιγάντιας πρόκλησης της ενεργείας των νέων. Πολλοί νέοι υπάρχουν ακόμα, οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο υπερβολικά νωρίς και οι τεράστιες δημοσιονομικές ε, περικοπές, η λιτότητα επίσης επηρεάζουν τους νέους. Εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στην κινητικότητα των νέων από περιφέρεια σε περιφέρεια και από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια πιο σωστά διατυπωμένη στρατηγική, πιο εστιασμένη για το μέλλον, ώστε να επικεντρωθούμε συγκεκριμένα σε αποτελεσματικά μέτρα για την απασχόληση των νέων. Τρία πράγματα θα ήθελα να επισημάνω. Το πρώτο είναι η εγγύηση της απασχόλησης. Διότι γνωρίζουμε ότι όταν ένας νέος παραμένει άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται όλο και πιο απίθανο να βρει κάποτε απασχόληση. Κατά συνέπεια πρέπει να βελτιώσουμε τη μετάβαση από τη φάση εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι κανένας δεν θα πέσει στα κενά μεταξύ των δύο. Και επίσης πρέπει να αυξήσουμε το διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργοδοτών ώστε να συμφωνούν οι δεξιότητες των ατόμων που παίρνουν κάποιο πτυχίο, κάποιο χαρτί με τις απαιτήσει της αγοράς. Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την αγορά εργασία. Έχουμε προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω το Εράσμο και το Νταβίντσι που βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και γλωσσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν για την πρόσβαση στην απασχόληση στη χώρα τους και αλλού. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τους νέους που υποστηρίξαμε, εγκρίναμε εδώ στο Κοινοβούλιο, υπάρχει για να ε, φροντίζει ώστε οι νέοι να βρίσκουν κάποια προσφορά απασχόλησης εντός μηνών αφού ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους ή αφού χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι σημαίνει ότι έτσι δεν θα χάνουν πάσα ελπίδα οι νέοι να βρουν κάποια δουλειά. Το, ένα σημαντικό κομμάτι από όλα αυτά είναι η ορατότητα, η προβολή οι νέοι για να βρουν δουλειά πρέπει να είναι ορατοί, πρέπει να είναι ορατοί. Ε, ε, πρέπει και εμεί να, να, να προβληθούμε στου νέου. πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Twitter, το Facebook, πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα του. Χρειάζεται να του ενημερώνουμε περισσότερο για τα προγράμματα που υπάρχουν. Δεύτερον, χρειάζεται να συνεργασία, χρειαζόμαστε διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Πρέπει επίσης να εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές, τις βέλτιστες πρακτικέ κοιτώντα τι γίνεται σε χώρε με χαμηλή ανεργία των νέων. Ε, φυσικά τα κράτη-μέλη θα παίξουν κεντρικό ρόλο, καθώ και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι στην αγορά εργασία θα μπορούσαν να συμμετέχουν για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε μια συζήτηση με τους βουλευτές από το Εθνικά Κοινοβούλιο για να δούμε πώς θα βρούμε ένα πολιτικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι το μέλλον εξαρτάται από τους νέους. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για ένα μέλλον με ευημερία, ανάπτυξη και κοινωνική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχω τώρα για τη συζήτηση που έχουν ζητήσει το λόγο επτά ομιλητές Μπορούμε λοιπόν μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας να έχουμε μια καλή συζήτηση. Θα δώσω τρία λεφτά σε κάθε ομιλητή και παραμένει κάποιο περιθώριο για περαιτέρω συζήτηση ή ενδεχομένως για άλλους ομιλητές ή τουλάχιστον κάποια συζήτηση με τους ε, εισηγητές μας. Ξεκινά με τον κύριο Μπάκερ από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο που είναι μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών της ε, Ολλανδικής Γερουσίας. Αν ήσασταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήσασταν στην Ομάδα των Φιλελευθέρων, παρόλα αυτά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ομιλίες των εισηγητών. Πραγματικά είναι ανησυχητική κατάσταση σε ορισμένε χώρες. Εγώ στην Ολλανδία έχω τύχει να ζω σε μια χώρα που η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή. Ζω και εργάζομαι λοιπόν σε αυτή τη χώρα και ίσως έχω ορισμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν. Υπάρχει, παρά το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, ε, άνεση κατανομή τη εργασίας. Για παράδειγμα, οι νέοι με μεταναστευτικό παρελθόν έχουν δυσκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Μετά υπάρχει έλλειψη τεχνικού προσωπικού. Αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να αλλάξουμε την εκπαίδευση. Πρέπει να αποφύγουμε την εγκατάλειψη του σχολείου. Και αυτό είναι ένα από του πιο αποτελεσματικού τρόπου να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε εργοδότε και συνεργασία με εργοδότε οι οποίοι έχουν ανάγκη υπαλλήλων, προσωπικού και θα είναι σε θέση να επενδύσουν μαζί με την κυβέρνηση σε ορισμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Και θα εκπαιδεύσουν τους νέους για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας τις οποίες χρειάζονται. Αλλά πολύ περισσότερο σημαντικό από αυτό, από την εγγύηση ε, έβρεσης εργασίας, είναι η εγγύηση πρόσβασης στην αναζήτηση εργασίας. Μετά, να πω ότι σε όλες τις συστάσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, ξέρω ότι αυτό ίσως να μην είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά σας, είναι η μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και από τη δική μου εμπειρία στην Ολλανδία έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμα διότι η αγορά εργασίας προστατεύει τους ε, ηλικιωμένους και τους ε, σημερινούς εργαζόμενους. Έπειτα, Ίσως είμαι εκτός ε, θέματος, όμως δεν θέλω να πω ότι οι θέσει εργασία δημιουργούνται από την πραγματική οικονομία και κάτι που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο Κοινοβούλιο είναι σενάρια ανάπτυξη για την Ευρώπη. Και αυτό προποθέτει δημιουργία θέσεων εργασία στην πραγματική οικονομία. Και να επισημάνω την, ε, τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, οι οποίες είναι κάτι που πρέπει να ε, επαναδιαπραγματευτούμε με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Από ό,τι γνωρίζω, η Ιρλανδική Προεδρία έχει ως, στόχο της, ε, ως έναν από τους στόχους της ε, αυτών Και ο στόχος επίσης είναι 2% αύξηση για ανάπτυξη του ΑΕΠ. Και πιστεύω πως και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη και να ενεργοποιήσουμε την Κομισιόν να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις συγκεκριμένες σας προτάσεις. Και οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη από όλους αυτούς οι οποίοι εκπονούν συγκεκριμένα προγράμματα. Για την ε, Bundesrat τώρα έχει το λόγο η κυρία Μαργίτε Κον από την ε, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η οποία είναι στην Σοσιαλιστική και Σοσιαλδημοκρατική Πτέρυγα. Έχετε το λόγο κυρία Κόνραντ. κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της εγγύησης ε, για τους, ε, νέων, για τους νέους. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ που το συζητούμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πιστεύω πως ε, λίγα θέματα είναι τόσο σημαντικά και τόσο επίκαιρα και πρέπει να συζητηθούν και να υπάρξει στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια όσο αυτό το θέμα. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε ε, παρατηρήσεις. Είμαι μέλος ε, της Επιτροπής αυτής στο Bundesrat και πιστεύω ότι αυτό το θέμα ανήκει πολύ περισσότερο σε αυτήν ε, την Επιτροπή. Είναι αντικείμενο έντονων συζητήσεων, είναι πολύ επίκαιρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, για την ε, πολιτική εξυγίαση των δημοσιονομικών. Πιστεύω πως δεν είναι εύκολο θέμα να λυθεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την στενή συνεργασία, αυτή την ενασχόληση με αυτά τα θεμελιώδους σημασίας θέματα. Και πιστεύω πως από τη στιγμή που αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι πολιτικοί κάνουν το ίδιο, οικονομία, λιτότητα, ότι όσο το κάνουν αυτό δεν θα δημιουργηθεί καμία προοπτική ανάκαμψης. Και το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Όσον αφορά τον, ε, τις εγγύησεις για τους νέους εντυπωσιάστηκα από τις εκθέσεις που μόλις άκουσα και από αυτό πιστεύω πως ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς, αυτό που συνδέει. Τι είναι αυτό που συνδέει. Οι επιπτώσεις της έλλειψης προοπτικής στους νέους. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλους μας, που θα επηρεάσει όλους μας και θέλω όλοι να ασχοληθούμε και να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Ποιες είναι οι προοπτικές και, ποια είναι το ποσοστό, και ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να κάνουμε προεκλογική εκστρατεία στην Ευρώπη, να κάνουμε πολιτική χωρίς να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Τι θα πούμε στους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους λέμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την ε, ενιαία αγορά, να ενοποιηθούν τα δημοσιονομικά, να σώσουμε τις τράπεζες. Αυτό που μπορούμε να εξηγήσουμε πολύ απλά στους ανθρώπους είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες τους. Πώς θα βελτιώσουμε την ζωή τους στην Ευρώπη και όχι πώς θα την επιδεινώσουμε. Και μόλις όλοι οι πολιτικοί ασχοληθούν με αυτό το βασικό ερώτημα, τότε μπορώ να πω ότι θα έχουμε πάει παραπέρα. Χρειαζόμαστε εγγυήσει για του νέου και σε αυτό το σημείο να δώσω άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, για αυτήν την συνεργασία. Και να κλείσω με τις ευχαριστίες μου και να αναφέρω ότι και αυτό ερώτημα δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και το τι γίνεται στα επιμέρους κράτη-μέλη. Τι κάνει κάθε κράτος μέλος για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Και αυτό είναι ένα θέμα που ανήκει σε κάθε σύνοδο κορυφής. Είναι εξίσου σημαντικό όπως όλα τα άλλα ερωτήματα, όπως οι εκθέσεις για την ανάπτυξη. Και πιστεύω πως μαζί, πως με συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Τώρα τα προγράμματα που αναφέρετε, να πω ότι είναι πολύ χρήσιμα, ιδιαίτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αναφέρατε και αυτό το υποστηρίζω απόλυτα. Η δομή όμως της ανεργίας των νέων διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα και γι' αυτό θα ήθελα εδώ να ζητήσω την πανευρωπαϊκή υποστήριξη σε μια μεγάλη ευελιξία εφαρμογής των προγραμμάτων, διότι τα προγράμματα πρέπει να προσαρμοστούν αναχώρα είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, προποθέσει, πολύ διαφορετικό background από χώρα σε χώρα. Και τέλος το ζήτημα της χρηματοδότησης. Πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο της χρηματοδότησης. Και το λέω αυτό ω Γερμανίδα και ξέρετε στη χώρα μου τώρα στο Κοινοβούλιο γίνονται συζητήσεις για περικοπές στον προϋπολογισμό. Όμως πιστεύω ότι αυτό εδώ πρέπει να ενισχυθεί. Σας παρακαλώ, ας μην συζητούμε μόνο για το ESF. Είναι, είναι πολύ σημαντικό, αλήθεια. Είναι αναγκαίο όμως για τις συνθήκες τώρα να δούμε και έξω από αυτό. Δεν φτάνει το ESF για να λύσει το πρόβλημα. Ας μην έχουμε στο επίκεντρο μόνο αυτό λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι έτσι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω η η Γερμανίδα υπουργό ε, κατά την ΕΠΣΚΟ να κάνει παρόμοιες ε, προτάσεις. Έχουμε τον Αλεχάνδρο Σέρκας, ε, ευρωβουλευτή, εκτός από ευρωβουλευτής, είναι επίσης Ισπανός και μέλος της ομάδας των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Ένα για κάθε ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και είμαι πεπισμένος ότι και στις δύο πλευρές η συνεργασία μεταξύ μας σε, αυτή την, σε αυτές τις ημερίδες μεταξύ Ευρωπαίων βουλευτών και Εθνικών βουλευτών θα είναι ιδιαίτερα εμπλουτιστική και για τις δύο πλευρές. Ξέρετε ότι και εγώ ήμουνα για πολλά χρόνια βουλευτής στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι έχουμε μια χρυσή ευκαιρία με αυτή την πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία αυτή για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είναι μετριοπαθής, είναι περιορισμένη, είναι πιο περιορισμένη από αυτό που θα ελπίζαμε. Αλλά <clears throat> παρόλα αυτά έχουμε μια ευκαιρία για να αλλάξουμε μια κατάσταση η οποία είναι ικτρή. Η πρόταση αυτή βέβαια είναι περιορισμένη γιατί δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή εγγύηση. Την αφήνουμε στα χέρια των κρατών μελών που δεν έχουν πρόσθετους πόρους για να την υλοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που υπάρχουν και υπάρχει μια μεγαλύτερη υποχρέωση από την πλευρά των κρατών μελών. <clears throat> και δεν αφορά μονάχα τις κυβερνήσεις, αφορά όλους στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η απασχόληση είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί και θα λυθεί ως πρόβλημα όταν οι αγορές ανακάμψουν. Πρέπει να τα δούμε τα πράγματα με πιο ευρύ πνεύμα. Και ξέρω ότι αυτό το οποίο είναι στη χώρα μας είναι απλώς σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν οι συστάσεις προς την Ισπανία του 2011-2012 από το Συμβούλιο, που ουσιαστικά αντιγράφηκαν από τον ένα χρόνο στον άλλο. Παραγωγή χάρη η αίτηση να υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουν το ίδιο ακριβώς χαρακτήρα. Δεν μιλάνε ποτέ για την ενεργεία, δεν μιλάνε ποτέ για την ενεργεία των νέων αυτές οι συστάσεις. Αυτό σα δείχνει το επίπεδο ευαισθησία με το οποίο αντιμετωπίζει το Συμβούλιο αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικά μια τραγωδία για μια χώρα όπω είναι η Ισπανία. Γι' αυτό <clears throat> πιστεύω ότι πρέπει ω Εθνικά Κοινοβούλια και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά το θέμα αυτό, ώστε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τι δεσμεύσει που θα αναλάβουν και να είναι πραγματικέ αυτέ οι δεσμεύσει, να μην παραμείνουν στο επίπεδο ρητορική και μόνο. Και για το δεύτερο θέμα τώρα, για τι κοινωνικέ συνέπειε τη κρίση. Πιστεύω ότι είναι σαφές το δράμα εκατομμυρίων ατόμων που έχουν χάσει τις θέσεις εργασίες τους, χάνουν σιγά σιγά τα αγαθά τους, το σπίτι τους κτλ. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο είναι ίσως λιγότερο ορατό. Δεν είναι μονάχα τα ατομικά δράματα, είναι και τα συλλογικά δράματα. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποχρεώνει να ανατρέψουμε βασικά στοιχεία των συλλογικών συμβάσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το σύστημα κοινωνικής ε, κάλυψης, το υγειονομικό σύστημα. Υπάρχει εκμετάλλευση της κρίσης για να εξαλειφθούν βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που εναπόκειται ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια να αγωνιστούν για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να υψώσουν τη φωνή τους γιατί όπως και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η Κομισιόν δεν είναι εδώ για να υποστηρίξει μόνο τις αγορές, είναι εδώ για να υποστηρίξει το κοινωνικό υπόδειγμα της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να προωθεί την καταστροφή των κοινωνικών προτύπων, θα πρέπει αντίθετα να διαφυλάξει αυτό το κοινωνικό πρότυπο και εδώ μπορούν να συμβάλλουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε στα Εθνικά Κοινοβούλια με τον συνάδελφό μας κύριο Γεροντοπλό που είναι υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκ μέρου του ΕΛΚ μάλιστα, Νέα Δημοκρατία. Έχετε αγαπητέ συνάδελφε το λόγο για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, προέρχομαι από την Ελλάδα, μια χώρα που βρέθηκε στο κέντρο της κρίσης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα βρισκόμαστε ως χώρα σε καλό δρόμο με μεγάλες θυσίες από τον ελληνικό λαό και με την ανεργία κυρίως των νέων να καλπάζει. Όπως ανέφερε προηγουμένως και ο κ. Κρεμαστινός, στους νέους μεταξύ 15-25 ετών η ανεργία είναι περίπου 57%. Όμως η κρίση στην Ευρώπη ήταν προβλέψιμη. Γιατί? Διότι ε, στην, στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση υπήρξε ένα προθύστερο, ένα πολιτικό παράδοξο. Προχωρήσαμε στην νομισματική ενοποίηση χωρίς χρόνος να έχουμε οικονομική τραπεζική και δημοσιονομική ενοποίηση. Και βεβαίως χωρίς να έχει προηγηθεί η πολιτική ένωση με κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Θα ήθελα να ρωτήσω, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ουσιαστική ενοποίηση της Ευρώπης. Χάσαμε την ευκαιρία στη Λισαβόνα, όπου φοβηθήκαμε να εκπονήσουμε ένα κοινό σύνταγμα, να μην χάσουμε και την ευκαιρία που μας δίνει η σημερινή κρίση έστω και αν κάποιες χώρες αποφασίσουν να μην ακολουθήσουν. Και επειδή το θέμα της συζήτησης είναι η ανεργία, θα ήθελα να αναφέρω μια βασική αιτία. Οι γειτονικέ χώρες, όπως ανέφερε και το πρωί ο συνάδελφος από την Λιθουανία, έχουν πολλές φορές δημιουργήσει φορολογικούς παραδείσους με φτηνά εργατικά χέρια. Τι πρέπει να γίνει. Καταρχάς η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της περιφέρειας της Ευρώπης αποτελεί τη μόνη λύση. Κάτι που θα ωφελήσει και τις ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζονται επίσης να δημιουργηθούν προγράμματα νεανικών επιχειρήσεων που θα συνοδεύονται με φοροαπαλλαγές για τους νέους ανθρώπους που επενδύουν. Και βεβαίως η Ευρώπη μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει και προγράμματα εκπαίδευσης ανέργων σε τομείς παραγωγικούς, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες, ο τουρισμός και η γεωργία. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη και οι χώρες μας ε, οφείλουν να προσφέρουν στους ανθρώπους τέσσερα βασικά αγαθά. Παιδεία, υγεία, ασφάλεια και βεβαίως εργασία. Εάν αυτά τα πράγματα δεν τα προσφέρουν, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής τους. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σούτς. Βελσκζίν, μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλή των Αντιπροσώπων των Κατοχωρών. Μέλος της ομάδας που εδώ στους φιλελεύθερους. Έχετε τρία λεπτά. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, οι 100 χώρες έχουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ενέργειας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιώθουμε πολύ άσχημα που βλέπουμε να είναι το πρώτο πράγμα που ανεβαίνει σε, περιοχή, σε εποχές η ανεργία των νέων. Η ύφεση είναι η αιτία για όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε γενικά μέτρα για να τονώσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση και να κρατήσουμε χαμηλά την ενεργεία. Αυτό θα ωφελήσει όλους όσους χρειάζονται δουλειά. Η Ολλανδική κυβέρνηση αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εγγύηση των Νέων, διότι εταιρείε δημιουργούν θέσει εργασία. Εμεί προσπαθούμε να τι δημιουργήσουμε τεχνητά και αυτό δεν είναι θετικό. Αυτέ οι δουλειέ δεν θα είναι βιώσιμε θα μειωθούν μόλις σταματήσουν οι επιχορηγήσεις. Όπως δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία, εμείς πιστεύουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένο ρόλο να παίξει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Και άλλοι ευρωβουλευτές ε, μας ζήτησαν να μάθουν τις βέλτιστες πρακτικές στις κατοχώρες. Έχουμε ένα μείγμα των δύο. και το μαστίγιο και το καρότο. Ένα συνδυασμό των δύο. Αυτό υπήρξε το πιο επιτυχές μέτρο μέχρι στιγμής. Χρησιμοποιήθηκε ως γενική πρακτική βάσει της νομοθεσίας. Δεύτερον, τα κίνητρα, το καρότο δηλαδή, η εργασία, η εκμάθηση για 16χρονους, 17χρονους που είναι μαθητές και δουλεύουν για λιγότερο από 16 ώρες την εβδομάδα. Αν είναι άνω των 18 και εξακολουθούν να σπουδάζουν, τους παρέχουν κάποια ωφέλη, του παρέχει κάποια ωφέλη η κυβέρνηση. Τρίτον, προσπαθούμε να συνδέσουμε την εκπαίδευση και τις αγορές εργασία σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση και ε, τα ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση που να ζητείται από την αγορά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια συμφωνία μεταξύ ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργοδοτών δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την εργασία αυτή αυτή στις κάτω Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να καταφέρουμε να διατηρούμε χαμηλά την ανεργία. Για να ολοκληρώσω ως κρατημέλη θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο επίπεδο στο οποίο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Θα ήθελα να ακούσω τις εμπειρίες άλλων κοινοβουλίων με επιτυχείς εθνικές πολιτικές καταπολέμησης της ενεργείας των νέων. Με ποιο τρόπο το πέτυχαν αυτοί. Εμείς πιστεύουμε ότι οι εγγύσει για τους νέους δεν θα δώσουν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. με των προνομίων της Προέδρου για να σας πω ότι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πρόσφατο ψήφισμα, δεν λέμε ότι αυτή η εγγύηση είναι εγγύηση εργασίας. Δεν υπάρχει υποχρέωση να δημιουργήσουμε εκ του μηδανός θέσεις εργασίας. Το σύνολο αυτών των μέτρων <clears throat> που αναφέρατε ως μέτρα που ήδη υπάρχουν στις κάτω χώρες είναι ακριβώς αυτά που εγγράφονται στο πνεύμα της εγγύησης για τον νέον όπως την έχει παρουσιάσει και η Κομισιόν και που ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν στις 18 Φεβρουαρίου από τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συζήτηση σε λανθασμένη βάση. Θα επανέλθουμε πάντως στο τέλος της συζήτησης. Έρχομαι τώρα σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής Απασχόλησης, την Ινιές Ζουμπέρ, που έρχεται από την Πορτογαλία και είναι από την Ευρωπαϊκή ε, Ενωτική Αριστερά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ να θίξω ένα θέμα. και να έχω ενδεχομένως και τα σχόλια των ε, ομιλητών μας, των εισηγητών μας και ιδίως από την πλευρά της εκπροσώπου του Φιλανδικού Κοινοβουλίου που νομίζω ότι είναι ήταν η πιο συγκεκριμένη παρέμβασή της σε σχέση με το μηχανισμό που θα μπορούσε να λειτουργήσει για την εγγύηση των νέων. Ένα από τα προβλήματα τα πιο έντονα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι πέραν της ανεργίας είναι η επισφάλεια των συμβάσεων εργασίας. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα σταθερότητας, είναι, δεν έχουν σταθερότητα στη ζωή τους, δεν έχουν τρόπο να σχεδιάσουν τη ζωή τους, δεν έχουν τα, τα δικαιώματα στον χώρο εργασίας που είχαν οι προηγούμενες γενιές και που τώρα χάνονται. Είναι συγχρόνως όμως και ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με την ε, δημιουργία υψηλότερου ή χαμηλότερου επίπεδου εργαζομένων. Γιατί ξέρουμε ότι η επισφαλής εργασία είναι ο προθάλαμος της ανεργίας. Όποιος μπαίνει σε μια τέτοια σχέση εργασίας ξέρει ότι αργά ή γρήγορα θα μπορέσει να απολυθεί πολύ εύκολα. Κατά την άποψή μου λοιπόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε και τις συμβάσεις εργασίας που έχουν επισφαλή χαρακτήρα. Για, τις, ε, για τα στάσια για τις ε, δράσεις μαθητείας. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση αυτών των στάζ με κάποια σύμβαση εργασίας. Και το επόμενο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι διαδικασίες μαθητείας, τα στάζ συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεν αντικαθιστούν εργαζόμενους, μόνιμους εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν αυτές τις θέσεις και επομένω είναι θέσει οι οποίε θα πρέπει να καλυπτόντουσαν με μια κανονική σχέση εργασία. Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με την υποστήριξη που δίνεται στου ε, εργοδότε. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μια υποστήριξη για το μισθολογικό κόστος 100 ευρώ το μήνα για τις ε, θέσει αυτές εργασία για νέους εργαζόμενου. Εδώ πέρα το ερώτημα μου το εξή. Υπάρχει κάποια, κάποιος υποχρεωτικός χαρακτήρας για τις ε, σχέσεις αυτές εργασίες, δηλαδή υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη μετά από το τέλος της περίοδου μαθητείας που υποστηρίζεται ή της εργασίας που υποστηρίζεται από αυτή την επιδότηση να προσλάβουν πραγματικά κάποιους εργαζόμενους γιατί ο κίνδυνος είναι αυτές οι επιδοτήσεις να τύχουν εκμετάλλευσης από τους εργοδότες οι οποίοι παίρνουν κόσμο, τον απολύουν και παίρνουν νέο κόσμο πάλι με την επιδότηση αυτή αντί να καλύπτουν αυτές τις θέσεις με συμβάσεις αόριστου χρόνου. Δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων τώρα, ο κύριος Άξελ Σέφα και η κυρία Μαρία Πλάτς. Ο Άξελ Σέφερ τον γνωρίζετε, υπήρχε υπήρξε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1994 στο 1999. Είστε αντιπρόεδρος ομάδος S5 στην ε, Bundestag και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσει Καταρχά, θεωρώ πολύ καλό το γεγονό ότι ε, ψηφίστηκε αυτή η έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την απέτηση για, για τι εγγύσει ε, για του νέου. Ε, πιστεύω πω και εμεί στα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να αναλάβουμε τι ίδιε δεσμεύσει. Και για αυτήν την έκθεση, όπως και για άλλες σημαντικέ εκθέσει αντίστοιχε. Πιστεύω πως αυτή είναι η καλύτερη και πιο αποδοτική μορφή συνεργασίας και για το μέλλον άλλωστε. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω. Είμαι υπέρ της παροχής εγγυήσεων και υπέρ του να πολεμήσουμε γι' αυτό. Χρειαζόμαστε υπεύθυνη πολιτική και η υπεύθυνη πολιτική έχει άμεση σύνδεση με το κράτος και με εγγυήσεις. Δηλαδή χρειαζόμαστε και κρατικές εγγυήσεις εάν θέλουμε εγγυήσεις για τους νέους. Ιδιαίτερα σε τέτοια, τέτοιες δραματικές περίοδους που διανύουμε. Τρίτον, στις αρχές της χιλιετίας η Γερμανία θεωρούταν ο ασθενής της Ευρώπης. Κάναμε βαθιές δομικές μεταρρυθμίσεις και αυτό κόστισε και στον ε, καγκελάριο Σρέντερ τη θέση του. Και τώρα η καγκελάριος ναι. Μέρκελ βρέπει τις Δάφνες αυτών των πολιτικών των σοσιαλιστών. Από τη μία έπρεπε να εξοικονομήσουμε και από την άλλη να επενδύσουμε εκεί όπου ήταν αναγκαίο. Και τρίτον, να διεξαχθεί και αυτή η δομική αλλαγή. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Πρέπει και τώρα να συνεχίσουμε να τα κάνουμε, εάν θέλουμε να αποφύγουμε αυτόν, αυτή τον κατήφορο. Και τέταρτον, θα ήθελα αυτό να το συζητήσω μαζί σας. Ως πρώην μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει κάποιοι αγώνες να γίνονται, να μεταφέρονται και θα το επαναλάβω, θα το θεωρούσα εξαιρετικά καλό, εάν το Κοινοβούλιο στη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο ασκήσει κριτική αν αυτό δεν είναι σωστό. Αν πει όχι, δεν συμφωνούμε και αν το κάνουν αυτό και τα άλλα ε, εθνικά κοινοβούλια, αν οι συνθήκε και οι διατάξει δεν είναι οι καλές, δεν είναι οι σωστέ, Και να τονίσω επίσης και τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στο δεύτερο τμήμα των εργασιών μας κυρίως όταν η κυρία Λόπε Φανθανιέ θα παρουσιάσει την εργασία της, διότι είναι ένα από τα θέματα που έχουμε στο πρόγραμμα και έχουμε εξετάσει για πολύ καιρό. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαρία Πλάτς και στη συνέχεια η κυρία Κορνέλισεν προετοιμάζεται. Κυρία Πλάτς, είστε μέλο τη Επιτροπής τη Αγορά Εργασία στη Σουηδία. Και εδώ θα ήσασταν μέλος της ομάδας του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσω τη σύσταση για την εγγύηση για τους νέους. Στο δεδομένο των υψηλών ποσοστών ανέργειας των νέων στην Ευρώπη. Αποτελεί θετική ένδειξη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζει η Κομισιόν έναν τρόπο εξόδου από αυτή την κρίση και μια κατευθυντήρια γραμμή για την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η σύσταση προσφέρει επαρκή ελαστικότητα ώστε να προσαρμοστεί εγγύηση στα συστήματα των διαφορών κρατών μελών και στους πόρους που είναι διαθέσιμους εκεί. Αλλά επίσης πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει ένα σαφές, ένα ηχηρό μήνυμα για το πόσο σπουδαία είναι η πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Στη Σουηδία θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση δεν πρέπει να ε, υπονομευτεί καθόλου, να μην ελαφρύνει καθόλου. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση της εγγύησης για τους νέους και στα κράτη-μέλη στο ήδη υπαρχόν πλαίσιο. Ταυτόχρονα χρειάζεται να σεβαστούμε το ρόλο των διαφορών κοινωνικών εταιρών στην αγορά εργασίας και το ρόλο του κοινωνικού διάλογου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καθαρή σας θέση. Ερχόμαστε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά θα επιστρέψουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια με τον Γοζενέρη. Προς το παρόν η κυρία Κορνέλισεν, μέλος των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προέρχεται από τις κατοχώρες. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Σήμερα κάθομαι με τους σοσιαλδημοκράτες. Είναι μια ευκαιρία για μένα. Δεν θα ήθελα να σταθώ τόσο στο περιεχόμενο αλλά στο θέμα της ε, δημοκρατικής νομιμοποίησης. Όπως γίνεται πολλές φορές με τις πολιτικές για τους νέους, δεν εμπλέκονται οι νέοι στις χώρες μας και το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν εμπλέκει τους νέους, αλλά βέβαια δεν εμπλέκει ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε την, ε, Τεχνικά Κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών κτλ. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά γενικά ισχύει αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, ώστε και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πλευρά του Εθνικών Κοινοβουλίων να τονίσουμε ορισμένα σημεία. Και εδώ θέλω να κάνω τρεις σύντομε προτάσεις για θέματα τα οποία και εμείς θα αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο άμεσο μέλλον. Το πρώτο θέμα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει εφέτος να υποβάλουν σχέδια για την απασχόληση με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους. Όλα τα κράτη-μέλη είχαν υποσχεθεί να το κάνουν αυτό στις 31 Ιανουαρίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2012 δεν έχουν τηρήσει αυτή την υπόσχεση. Θα είναι πολύ θετικό αν ζητήσετε και επιμείνετε να καταθέσει κάθε χώρα ένα εθνικό σχέδιο απασχόλησης και επίσης να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη πρόταση όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις των νέων στη συζήτηση για τα εθνικά πρόγραμμα τα απασχόλησης και στη συζήτηση για τις καταχώρα συστάσεις. Θα πρέπει να ζητήσετε από τις κυβερνήσεις σας να καταρτήσουν ένα σχέδιο για διαβουλεύσεις ή αν δεν το κάνουν αυτό να αργώνεστε εσείς κάτι κοινοβούλιο, εθνικό κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Και έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο Πολλές φορές οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια σε εθνικό επίπεδο οργανώνουν πολλές δραστηριότητες, κάποιες τις οποίες είναι καινοτόμε για τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Οι Γάλλοι είχαν μια στογγυλή τράπεζα, οι Βέλγοι κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν και θα ήταν χρήσιμο αν οι γραμματείες των Εθνικών Κοινοβουλίων να μπορέσουν να ανταλλάξουν πρακτικές και απόψεις για όλους αυτούς τους τρόπους με, τον, με τους οποίους τα κοινοβούλια μπορούν να εμπλέξουν τους νέους στην κοινωνία των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε λίγη περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Ξαναγυρίζω στα Εθνικά Κοινοβούλια με τον Ρώσο Ενεγκρή από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες του Λουξεμβούργου. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έπρεπε να αναπτύξουμε περισσότερο σε μεγαλύτερη κλίμακα την αλληλέγγυα οικονομία για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Η κοινωνική οικονομία επίσης θα μπορούσε να προσφέρει στους νέους πρόσβαση, αν όχι άμεση, τουλάχιστον δεύτερο πυλώνα στην αγορά εργασίας. Αντί είναι να μένουν στο σπίτι και να υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το μίσο που θα ήταν ενδιαφέροντες για τους νέους ε, συνοπτικά η εγγύηση για τους νέους δεν θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να πηγαίνει παράλληλα με την αλληλέγγυα οικονομία εάν τα υπόλοιπα μέτρα και προγράμματα δεν καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος δεδομένη τη συζήτηση που γίνεται, περνάω στα πέντε μέλη του πάνελ για να ρωτήσω αν κάποιος από αυτού. θα ήθελε να μιλήσει για να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο την ανταλλαγή και να απαντήσουν στα όσα ακούσαμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα στα οποία θα θέλαμε να επανέλθουμε. Η κυρία Φιλατόβ ζήτησε το λόγο. Σα δίνω λοιπόν ευχαριστώ το λόγο. Καθώ γραφτήκατε πρώτοι, θα μιλήσετε πρώτοι. κάποιο άλλο κύριο Κρίστενσεν και εσείς. Εσείς ναι ή όχι, τώρα πρέπει να το πείτε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις λοιπόν. Δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για τα θέματα αυτά, αληθεύει το ότι οι βραχυχρόνιες σχέσεις εργασίας είναι μια μάστιγα για τους νέους, αλλά ακόμα και η βραχυχρόνια εργασία είναι καλύτερη από την ανεργία. Όταν υποστηρίζουμε την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, από τις επιχειρήσεις, ένα τμήμα αυτής της βοήθειας πηγαίνει και στις επιχειρήσεις κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ακόμα Και αν υπάρχει μεγάλη προσφορά θέσεων απασχόληση, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα των νέων. Πολλοί νέοι δεν θα μπορέσουν να έχουν θέσει εργασία γιατί δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, δεν έχουν τι ικανότητε και αυτέ οι κρατικέ βοήθειε δεν βοηθούν το άτομο να προχωρήσει στην επαγγελματική του καριέρα. Έχουμε συζητήσει για το πώ μπορούμε να περιλάβουμε καλύτερα του νέου στο χώρο εργασία στη Φινλανδία και να διευρύνουμε την οικίσια του νέου. Χρησιμοποίησαμε ιδιαίτερα το διαδίκτυο κάνοντας ε, συζητήσεις μέσα από το διαδίκτυο και ιδιαίτερα το facebook. Πώς λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες για τους νέους, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης και η πρόκληση για μας είναι να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και έτσι να ξέρουμε καλύτερα τι θέλουν και οι νέοι και όχι απλώς να επιβάλλουν οι πιο ενήλικες στους νέους, οι πιο ηλικιωμένοι στους νέους, τη δική τους άποψη για το πώς πρέπει να είναι ο νέος ή πώς σκεφτόντουσαν αυτή τη νεότητα όταν ήταν τότε εκείνοι οι νέοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και εδώ στέκομαι μονάχα στο θέμα της γενικής πολιτικής, πώς δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης, πώς ε, έχουμε ανάπτυξη αν δεν έχουμε αρκετή ε, προσφορά εργασία οι νέοι θα υποφέρουν περισσότερο. Ο Όλε Κρίστενσεν. Έχουμε ένα άριστο παράδειγμα λοιπόν από τη Φιλανδία. Δείχθηκε η γνώμη των νέων και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. ήθελα να κοιτάξουμε τις δύο απόψεις που ακούσαμε. Η εκπρόσωπος των κατοχωρών είπε ότι οι δημοσίες αρχές δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα ο συνάδελφος από το Λουξεμβούργο είπε ότι χρειαζόμαστε κάτι που να κρατά απασχολημένους τους νέους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα χρειαστεί να βρούμε μια ισορροπία. Πρέπει να διατηρούμε απασχολημένους τους νέους ώστε να μην χάσουμε πολλές γενιές. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια δημογραφική πρόκληση στην Ευρώπη Εάν δεν κρατήσουμε απασχολημένους τους νέους, θα τους χάσουμε στο μέλλον. Με έναν τέτοιο συνδυασμό, οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να διδρούν απασχολημένους τους νέους, ώστε να είναι έτοιμοι, να είναι χρήσιμοι στο μέλλον. δεν θα αρκέσουν οι επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δράσουν όλα τα κράτη-μέλη για να αποκομίσουμε τα ωφέλη των επενδύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο συνάδελφο ε, Άσπυρο Φίλαρ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσε όλε αυτέ τι ε, παρατηρήσει. Βέβαια κάθε χώρα έχει το δικό της ιστορικό, τη δική της παράδοση στα θέματα της απασχόλησης. Εγώ έρχομαι από τη χώρα των Βάσκων όπου η ανεργία είναι κατά το 1 τρίτο χαμηλότερη από την ε, ανεργία στην υπόλοιπη Ισπανία. Δεν υπάρχει λοιπόν μια ομοιογενής και ομοιόμορφη κατάσταση σε όλες τις χώρες. Βέβαια, όταν έχουμε φτάσει στο 55% ανεργία των νέων, είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ κατανοώ λοιπόν αυτά τα οποία ελέγχθησαν ότι πρέπει να γίνει κάτι και σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας. Αλλά τι είναι η πραγματική οικονομία. Όταν εγώ φτιάνω ένα αυτοκινητόδρομο, αυτό είναι κάτι που προέρχεται από την πραγματική οικονομία ή όχι, ή είναι κάτι το οποίο αποφασίζει κάποιος. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα ένα περιθώριο ελιγμών <clears throat> για την κρατική δράση, όπου θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Η Ισπανία, κύριε Θέπε, είναι σε κατάσταση εξυγίανσης των οικονομικών, όπω ξέρετε πολύ καλά, και γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειε προ την κατεύθυνση αυτή. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ δεν έχει τηρήσει τα υπεσχημένα στις εκλογές. Αναγκάζεται να αυξήσει τους φόρους παρά τη φιλοσοφία του. Θέλει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει η μείωση του ελλείμματος για να μπορέσουμε να είμαστε φερέγγοι και αξιόπιστη και να μπορούμε να αξίζουμε την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Γι' αυτό έχουμε μπει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα δώσουν κάποια δυνατότητα ανάκαμψης και επομένως ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αναφέρθηκε το θέμα της κοινωνικής εργασίας. Στη χώρα μου υπάρχουν πάνω από 300.000 που εργάζονται σε διάφορες συνεργατικές μορφές εργασίας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νεότεροι των 40 ετών. Επομένως υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για τους νέους στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Και εδώ θέλω να κάνω την εξή παρατήρηση. Η χρηματοπιστωτική κρίση είναι η πηγή όλων των κακών ελέγχθη. Σχεδόν, σχεδόν. Σίγουρα όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση είναι υποχρεωμένε οι επιχειρήσει να κλείσουν ή πολλέ φορέ πτωχεύουν οι πελάτε του, οι προμηθευτέ του και του οδηγούν σε δύσκολη κατάσταση. Όλα αυτά μα οδηγούν όμω στην εξή σκέψη. Είμαστε σε μια κατάσταση μεταλλαγή με την παγκοσμιοποίηση και τι νέε τεχνολογίε που αλλάζουν τη μορφή τη εργασία. Για τα δύο αυτά θέματα πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κρίστερσεν, ο οποίο μίλησε για κάτι για το οποίο εμεί δεν έχουμε αναφερθεί ιδιαίτερα. Το θέμα τη δημογραφική αλλαγή, το γεγονό ότι γυράσκει η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη δείχνει να μην έχει μέλλον. Είναι πολλέ χώρε, όπω και η δική μου, οι οποίε αυτοκτονούν σε δημογραφικό επίπεδο. Αυτό θα έχει μεγάλες Επιπτώσει στο κράτο ευμάρειας τη χώρα μα. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα, γιατί αν δεν υπάρξουν ενεργέ πολιτικέ υπέρ τη γεννητικότητα, θα υπάρχει πρόβλημα. Και οι πολιτικέ αυτέ θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να αποδώσουν καρπούς. Αν η Ευρώπη θέλει να έχει ένα μέλλον, θα πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην εισηγητριά μας ε, για την απασχόληση των νέων, την κυρία Στρίσλευσκα και μετά θα ακούσουμε τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως βλέπετε, η σημερινή συζήτηση τι μας έχει δείξει ότι χωρίς συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο να βελτιώσουμε την κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις ε, πολύ επικοδομητικές συνεισφορές σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, εκπρόσωπο από την Φιλανδία, διότι οι ιδέες που είχε μου πάρα πολύ. Δηλαδή η δεκάμινη απασχόληση κατά την οποία ο εργοδότης θα λαμβάνει 700 ευρώ για κάθε απασχολούμενο. Αυτή η ιδέα με βρίσκει πολύ σύμφωνη και πιστεύω ότι το θέμα του Youth Guarantee, το, της εγγύησης για τους νέους, πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά την Πρόεδρό μας κυρία Μπερές και να πω ότι ελπίζω να δημιουργήσουμε μία έκθεση η οποία δεν θα μείνει μόνο στα χαρτιά, αλλά θα αλλάξει πραγματικά την κατάσταση των νέων και στην αγορά εργασίας. Ελπίζω λοιπόν σε μια επικοδομητική συνεργασία και ελπίζω επίσης οι πολιτικές ε, ομάδες να έχουν καλή συνεργασία, να υπάρχει συνένεση, διότι πραγματικά πρέπει να συνεργαστούμε καλά και να φροντίσουμε να μην πάει χαμένη μια ολόκληρη γενιά. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω και αυτό που είπε η κυρία Ζούμπερ. Είπε πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια όταν κάποιος προσλαμβάνει έναν νέο. Πολλές φορές οι εργοδότες χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται το σύστημα και το υπονομεύουν με αυτόν τον τρόπο. Έχω προσωπική εμπειρία με αυτό το θέμα. Όταν ήμουν φοιτήτρια δούλευα σε μια εταιρεία και ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί. Όταν όλοι οι εργοδότες πρέπει να απασχολήσουν, θα είναι υποχρεωμένοι να απασχολήσουν έναν μαθητευόμενο, τότε η κατάσταση πιστεύω να αλλάξει προς το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ συμπερασματικά να κάνω έξι παρατηρήσει. Η πρώτη έχει ως εξή. Πιστεύω το ζήτημα της απασχόλησης των νέων ε, φέρνει στο νου αυτή την έννοια της χαμένης γενιάς. Κινητοποιείται λοιπόν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους στόχους βιωσιμότητας. Ε, Γαλλία λέμε, στη Γαλλία λέμε sustainability, για το sustainable, αυτή τη βιωσιμότητα. Το χρησιμοποιούσαμε καταρχάς για το περιβάλλον, αλλά πρώτα απ' όλα πιστεύω πριν το περιβάλλον θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τον ανθρώπινο παράγοντα να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο της χαμένης γενιάς που θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες απώλειες της κοινωνίας μας. Ε, μια κοινωνία που γυράσκει το ζήτημα λοιπόν αυτό, το να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ε, της ε, κινητοποίησης ε, είναι σημαντικό. Όταν λοιπόν οι μεγάλοι μας εμπειρογνώμονες λένε ότι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση είναι η καινοτομία, πάντα έτσι αναφέρεται πρώτη η καινοτομία. Αυτή είναι η σωστή οδός που πρέπει να ακούσουμε και ποιος άλλος εκτός από τους νέους είναι εκείνος που θα μπορούσε καλύτερα να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση της καινοτομία. Αυτοί έχουν νέες ιδέες. Οι νέοι έχουν ταλέντα και την ικανότητα να μπορούν να επιφέρουν καινοτομία. Ακόμη και αν δεν το κάνουμε από γενεοδορία, τουλάχιστον να το κάνουμε από εγωισμό. Αυτοί έχουν ικανότητα να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτή να ανακατανεμηθεί στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε τους νέους να δουλέψουν. Αυτό μας φέρνει στη δεύτερη μου παρατήρηση. Σχετίζεται με τα όσα είπε ο συνάδελφος Μπάκερ από τις κατοχώρες για, αφορά το να αποφύγουμε την πρόορια εγκατάλειψη του σχολείου. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ τι συμβαίνει με όσους είναι ανειδίκευτοι αφενός και της πρόκλησης που αυτός είναι πάγεται. Συζητούσα τις προάλλες με έναν επίτροπο και του μίλαγα για αυτά το ταλέντο των νέων, την ικανότητά τους να καινοτομήσουν και αυτός μου έλεγε «Μα δεν έχουν εξειδίκευση». Είναι χωρίς εξειδίκευση όμως διότι εμείς ε, δεν έχουμε συνδέσει σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα και την εξέβριση εργασίας. Όσοι είναι άνεργοι σήμερα δεν είναι απαραίτητα ανειδίκευτοι. Είχαμε πει στο ψηφισμά μας ότι θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε για τους νέους έως 30 ετών που είναι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ξέρω ότι συμβαίνει αυτό στην Ισπανία, αλλά όχι μόνο. Έχουμε νέους πτυχιούχους που ούτε αυτοί δεν βρίσκουν εργασία. Δεν είναι θέμα λοιπόν έλλειψης προσόντων είναι θέμα έλλειψη σύνδεση μεταξύ ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αγορά εργασία. Ε, θα ήθελα να επανέλθω και στα όσα είπε ο συνάδελφο ο κ. Κρεμαστινό και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ε, νούμερα τα οποία πήρα από τον Ζακ Ντελαροζιέρ, που τα γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Είναι ανησυχητικό. Όταν κοιτάμε την αγορά εργασία, σήμερα όσοι είναι εργάτες με ένα πτυχίο όχι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λιγότερο από αυτό και που έχουν εργασία στην ε, Γερμανία κατέχουν το 16% του εισόδου εργασίας. Το 16% δηλαδή των εργαζομένων, των εργατών στη Γερμανία έχουν ένα δίπλωμα επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή χαμηλότερο από το απολυτήριο. 70% είναι αυτός, ε, αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο στην Πορτογαλία. Το ζήτημα λοιπόν του διπλώματος, του, του απολυτηρίου είναι σημαντικό. Επίσης ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η κυρία Κορνέλισον για το διακύβευμα για τα κράτη-μέλη που έχουν αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη να παρέχουν σχέδια απασχόλησης. Είναι ζωτική σημασίας θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αποτελεί το επίκεντρο της συζήτησή μας. Αν πιστεύουμε σε, αυτή, την εκ σε αυτόν τον εκ των προτέρων συντονισμό και στο ότι πρέπει να θέσουμε την απασχόληση ως προτεραιότητα και αυτό συνάδει και με την παρατηρήση της κυρίας Κόντρα δεν αρκεί να σκεφτόμαστε να έχουμε στο νου μας επενδύσεις και ανάπτυξη. Πρέπει να θέλουμε να θέσουμε στο επίκεντρο το ζήτημα της απασχόλησης. Πρέπει κάθε κράτος μέλος να πει όχι μόνο πώς θα δημιουργήσει ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα της απασχόλησης. Στη συνέχεια, όταν η Κομισιόν ορίζει συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα, πρέπει να μην ε, επαναπάβεται με το πώς θα διοργανώσει τη δημοσιονομική πειθαρχία τα κράτη-μέλη, αλλά και με το πώς ε, θα καταφέρουν να επιτύχουν αυτή την ισορροπία που ανέφερε ο Αξεσέφερ που υπήρχε στις μεταρρυθμίσεις και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε όλα αυτά να καταλήξουν σε πραγματική δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό που κατάφερε ο Επιτρόπος Αντόρ κατά την ετήσια ανασκόψη φέτος όπου είπε ότι αυτό ο τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν το στόχο για του νέου στα κράτη-μέλη πρέπει να εντάσσεται στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Έτσι, ερχόμαστε στην τέταρτη μου παρατήρηση που σχετίζεται με την ε, παρατήρηση της, ε, του συναδελφού Κόντραντ ε, σε σχέση με τις στρατηγικές που δημιουργούν απασχόληση ή όχι. Οι συναδέλφοι ευρωβουλευτές το γνωρίζουν απ' έξω. Το λέω σχεδόν σε κάθε συνάντησή μας και του ζητώ συγγνώμη. Αλλά μια αντικειμενική παρακολούθηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ακόμη και πριν την κρίση, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι μια απλή στρατηγική απασχόλησης, ακόμη και επένδυσης υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, δεν θα αρκέσει αυτή καθεαυτή για να επιλύσει το ζήτημα της απασχόλησης. Ως απόδειξη μπορούμε να δούμε τα 10 χρόνια πριν την κρίση. Τότε είχαμε ανάπτυξη της τάξης του 2%. Και μα είχαν πει ότι αυτό ήταν το κατόφλιο δημιουργία θέσεων εργασία. Αλλά ακόμη και σε εκείνη την περίοδο δεν δημιουργήσαμε τον αριθμό θέσεων εργασία που χρειαζόμασταν. Υπό αυτέ τι συνθήκε λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μα έδωσε η συνθήκη τη Λισαβόνα και που δεν χρησιμοποιεί κανεί. Αναφέρομαι ειδικότερα στο άρθρο 9, το οποίο λέει ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί μια πολιτική, όποια και αν είναι αυτή, πρέπει να εξετάζει τις ικανότητες, την αποτελεσματικότητα, τι επιπτώσεις έχει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μελέτη αντικτύπου δεν σημαίνει απλά δημιουργία μιας ε, ε, μελέτης αντικτύπου για να ακολουθήσουμε τις συμβουλές ενός συμβουλευτικού γραφείου. Είναι πραγματικά να δούμε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Έτσι ερχόμαστε στην πέμπτη μου παρατήρηση. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Έχω ένα όνειρο, I have a dream, ότι όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με όσα έκαναν ορισμένα εθνικά κοινοβούλια με τη φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπου υπήρχαν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτέλεσε γέφυρα προς κάτι που συμβαίνει και στα εθνικά κοινοβούλια. Να σκεφτούμε αυτή την εγγύηση για τους νέους, το έχετε στη Φιλανδία. Κάτι γίνεται και στην Αυστρία, όπως γνωρίζω, και στο Λουξεμβούργο. Τώρα έρχεται και στη Γαλλία με αυτό το Συμβόλο Γενναιών. Αρχίζει και εγκαθιδρύεται σιγά σιγά στη χώρα μας, καθιερώνεται. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πρωτοβουλία σε κάθε κράτος μέλος για να υποστηρίξουμε αυτή την εγγύηση για τους νέους. Να ασκήσουμε επίση την κυβέρνηση και να βεβαιωθούμε ότι εξακολουθεί η εστίαση στην εφαρμογή αυτή τη εγγύηση για του νέου, στο να γίνει πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι και υπό την Ιρλανδική Προεδρία θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα από την συνάντηση ΕΠΣΚΟ. Το τελευταίο σημείο είναι ότι ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η Σουηδή συνάδελφος νομίζω το να μην μειώσουμε την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι είμαι πεπισμένη ότι αυτό που προτείνει η Κομισιόν είναι ένας εξαιρετικός συμβιβασμός, ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός. Συμβιβασμός δεν θα μπορούσαμε να πάμε και πιο πέρα, θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν αυτόματο μηχανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά την παρούσα στιγμή αυτό που έχουμε μπροστά μας πιστεύω θα μπορούσε να γίνει δεκτό από όλους. Συμπεριλαμβανομένων το τονίζω αυτής της ιδέας ότι η εγγύηση για τους νέους θα πρέπει να υλοποιείται εντός τεσσάρων μηνών μετά από την ε, θέση του νέου αυτού σε μια κατάσταση όπου χρειάζεται αυτή την εγγύηση. Το φιλανδικό παράδειγμα αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η έννοια των τεσσάρων μηνών. Εντό αυτών των τεσσάρων <coughs> μηνών πρέπει να πιάσουμε το νέο πριν χαθεί από την αγορά εργασία. Το λέω καθαρά και δυνατά, διότι στο Συμβούλιο μερικοί λένε θα μπορούσαμε να πούμε έξι μήνε. Όχι. Όταν μιλάμε για εγγύηση για του νέου, πρέπει να αναφερόμαστε σε τέσσερι μήνε, ούτε πέντε ούτε έξι. Πιστεύω ότι βάσει όλων αυτών μπορούμε να συνεχίσουμε να, τη συνεργασία μας και να, η όθηση που όλοι θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την προτεραιότητα να γίνει πραγματικότητα. Και όσοι ελέγχουν τα κονδύλια να λαμβάνουν υπόψη και τις ε, πολιτικές προτεραιότητες, τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι των εργασιών μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες μας εδώ, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωκοινοβουλίου μπορούμε πιστεύω να τους χειροκροτήσουμε. Και μετά θα τους ζητήσω να ε, εγκαταλείψουν την έδρα διότι χρειαζόμαστε να έρθουν εδώ το πάνελ για το δεύτερο κομμάτι των εργασιών μας που αφορά τον αντίκτυπο της κρίσης. Euh, Αν θέλετε μπορείτε να καθίσετε κιόλα μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή για να περάσουμε στο δεύτερο μας θέμα. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι κεφαλαίο του σημασίας. Ο κοινωνικός αντίκτυπος των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στις χώρες που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες. Το πάνελ μας εδώ απαρτίζεται από τρεις συναδέλφους, δύο από τα Εθνικά Κοινοβούλια, η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλειας και Απασχόλησης του, Πορτο... του ο πρόεδρος του... της Επιτροπής αυτής στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, κ. Καναβάρου, και επίσης ο αντιπρόεδρος Αβεγκαντά από το λεκτορικό Κοινοβούλιο, δεν το είπα σωστά, σίγουρα, και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Βερόνικα Λοπέ Φοντανιέ, η οποία ήταν η συγγήτρια για την ετήσια έκθεση οικονομικής ανάπτυξης. Δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς θα σας πενθυμίσω πόσο μεγάλη είναι η σημασία αυτής της προβληματικής, πόσο σημαντικό είναι αυτοί που ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποια συνένωση για τα θέματα αυτά, ιδίω σε μια στιγμή που οι οικονομολόγοι συζητούν ατερμόνως για την σημασία του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή για την οικονομική προσαρμογή και φαίνεται ότι ο πολλαπλασιαστής αυτός δεν είναι μονάχα ένας πολλαπλασιαστής στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον κοινωνικό τομέα ιδίω και οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης απασχόλησης. Περί αυτού πρόκειται. και όταν εξετάζει κανείς, όπως έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, την επίπτωση που έχουν όλα αυτά στο να βγαίνουν από τον κοινωνικό χώρο, να βγαίνουν από τον χώρο της εργασίας και να περνάνε στο επίπεδο του αποκλεισμού του κοινωνικού μεγάλε ομάδε του πληθυσμού, αυτό είναι κάτι το οποίο μα οδηγεί σε μεγάλη ανησυχία. Χωρί να καθυστερήσω λοιπόν, θα δώσω το λόγο στου τρει εμπειρογνώμονέ μα από τον κοινοβουλευτικό χώρο. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον Ζουζε Μανουέλ Καναβάρου για 10 λεπτά. Είσαστε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε και για τη διοργάνωση αυτή και θέλω να χαιρετήσω όλους αυτούς οι οποίοι είναι παρόντες στην αίθουσα και συμμετέχουν σε αυτές τις ημερίδες. Θα μιλήσω τώρα στα πορτογαλικά κοινωνικός αντίκτυπος των διαδικασιών δημοσιονομικής εξυγίανσης και ιδίως για την Πορτογαλία. Αυτό είναι μια πρόκληση που θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω, αλλά φυσικά μιλάω προσωπικά, εκφράζω μονάχα την προσωπική μου άποψη. Είμαι βουλευτή σε ένα από τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την τωρινή πορεία προσαρμογής στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά δεν θα είμαι ε, στο βαθμό μπορώ μεροληπτικός. Η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και φιλολογία για τα θέματα αυτά ε, είναι γνωστή, αλλά δεν υπάρχει πάντα η ίδια ε, κοινή γραμμή για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό τομέα. Η προσαρμογή στα οικονομικά και δημοσιονομικά είναι κάτι με μεγάλο πολιτικό κόστος. Το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε το 2011 η προηγούμενη κυβέρνηση Πορτογαλία με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν προέβλεπε μερικού γενικού δείκτε που κατάδειχναν τη γενική κατάσταση και τον αντίκτυπο για τον πληθυσμό. Και υπήρχε πλήρη επίγνωση του προβλήματο τότε. Η Πορτογαλία έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εξυγίανση του προπολογισμού τη. Υπήρξε και ε, αναγνώριση εκ των έξω για τι προσπάθειε αυτέ, είτε από του φορεί που μα υποστηρίζουν ε, σε δημοσιονομικό επίπεδο, και επίσης, αλλά και επίσης από τις χρηματαγορές. Η Πορτογαλία γνώρισε αναγνώριση για τις προσπάθειές της και ακολούθησε ένα πρόγραμμα λιτότητος, ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα που για πολλούς από εμά ήταν απαραίτητη αυτή η λιτότητα. Άλλοι θεωρούν ότι ξεπεράσαμε όμως και το επίπεδο της απαραίτητης λιτότητας. Στην Πορτογαλία σήμερα έχουμε μια ανεργία 5% ανώτερη από αυτή που ίσχυε πριν υπογραφεί το μνημόνιο και περίπου περίπου 8% σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων και 1,5% ανώτερη σε ό,τι αφορά την ανεργία μεγάλης διάρκειας, πάλι σε σύγκριση πάντη με το πρώτο τρίμηνο του 2011 όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα προσαρμογής για τα οικονομικά θέματα στην Πορτογαλία. Είναι σαφές ότι ξεπερνάμε λοιπόν τη γενική τάση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των χωρών του ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι ο πιο σημαντικό κοινωνικό δείκτη. Δείχνει ότι υπάρχει μια έλλειψη, μια μείωση του εισοδήματο των ατόμων, μια μείωση των δημοσίων ε, επιδοτήσεων και των δημοσίων δαπάνων γενικά. Είναι σαφέ ότι αυτό είναι μια σημαντική παράμετρο στη συζήτηση που κάνουμε. Η κυβέρνηση Πορτογαλίας προσπάθησε να υπάρξει συμφωνία με τους ε, κοινωνικού εταίρους στα θέματα τη εργασία. έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ε, αν εξαιρέσουμε μία μεγάλη ε, οργάνωση συνδικαλιστική, να υπάρξει συμφωνία. Εκτός λοιπόν από την αριστερή αυτή οργάνωση. Υπήρξαν πολλές λοιπόν αλλαγές στον εργασιακό κώδικα που υποστηρίχτηκαν και από την κυβέρνηση και από τη σοσιαλιστική ομάδα που είναι στην αντιπολίτευση. Αυτές είχαν, οι αλλαγές είχαν σαν στόχο να ενισχύσουν την δυνατότητα αναπροσαρμογής στον τομέα της ε, απασχόλησης και να δυναμ... να γίνει πιο δυναμική η διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης των εργαζομένων. Η Πορτογαλία έχει κάνει λοιπόν μια σειρά από πρωτοβουλίε για του νέου με την υποστήριξη των κοινωνικών, κοινωτικών πόρων για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσει, οι κρατικοί φορεί, οι φορεί οι οποίοι προωθούν επαγγελματική κατάρτιση και στάση των νέων που μπορούν να οδηγήσουν στην απασχόληση και επίση είχαμε μια πρόσφατη ε, πρωτοβουλία για του πιο ηλικιωμένου και με λιγότερα προσόντα ε, άνεργος μακράς διαρκείας. Για τον τομέα αυτό η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να έχει μια πιο στενή συνεργασία για να μπορέσει να απαλύνει τα αποτελέσματα της λιτότητας και της κρίσης. Επίσης έχουμε καθορίσει ένα σχέδιο κοινωνικής έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες οι πιο άμεσες του πληθυσμού και ιδίω των πιο ευαλώτων στρωμάτων του πληθυσμού που ζουν με συντάξεις που είναι στο όριο τη δυνατότητα επιβίωσης ή έχουν αποδοχέ κάτω από τον ελάχιστο εθνικό μισθό, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιο επίγουσε ανάγκε ατόμων που έχουν ανεπάρκεια τροφίμων <clears throat> ή ανεπάρκεια βασικών υπηρεσιών. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τη λιτότητα και τη διαδικασία προσέγγιση, Είναι η αύξηση του χρέου των νοικοκυριών και εδώ υπήρξε και μια νομοθεσία για την υποστήριξη προς τις οικογένειες αυτές να αναδιαπραγματευτούν τα χρέη του με τις τράπεζες. Είναι προβλήματα λοιπόν όπου πάντα υπήρξε μία αντιμετώπιση από το κράτος. Υπήρξε μία μείωση ε, σειρά από προβλήματα που θα προκύψουν σε κοινωνικό επίπεδο χάρη λόγω μάλλον αυτών των περικοπών του δημοσίου προϋπολογισμού. Έχουμε ένα σύνολο από πολιτικές δημόσιες οι οποίες προσπαθούν να απαλύνουν τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Κάποιες από αυτές είναι αυτές τις οποίες αναφέρω στο έγγραφό μου. Πέραν λοιπόν από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Πορτογαλίας, οι συμπατριώτες μου και εκεί είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη και ιδίως η αλληλεγγύη σε επίπεδο οικογένειας, η δράσεις αυτές έχουν σαν στόχο να τεθούν από κοινού η, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και να μειωθεί ο αντίκτυπος των προβλημάτων μας. Είμαστε μια μικρή κοινότητα, κοινωνία στην Πορτογαλία, αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μια μεγάλη μικρή κοινωνία. Απαρτιζόμαστε από μικρές κοινωνίες οι οποίες συνενώνται σε μια μεγάλη. Και οι Πορτογάλοι έχουν καταφέρει να αντισταθούν στην κρίση, να κάνουν πρωτοβουλίες και να διακρίνουν και δυνατότητες λύσεις για το μέλλον. Τα μακροοικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με λύσεις σε μικροοικονομικό επίπεδο. Αλλά είναι δυνατόν με μικρές προσπάθειες αυτού του είδους να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του κράτους μας. Και όλες αυτές οι προσπάθειες μας κάνουν να αξίζουμε περισσότερο την υποστήριξη των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μα Σάρβιλ Σαζερντέν, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση ε, του Λετωνικού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρωτού μιλήσω για την κατάσταση στην ε, Λετωνία και για τις λύσεις που έχουμε βρει, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο για την επιλογή του προηγούμενου θέματος που συζητήσαμε. Η θέση μας ε, ήταν πιο συντηρητική παλιότερα και νομίζω πως τώρα καταφέραμε με βάση αυτή τη συζήτηση να αλλάξουμε τις απόψεις μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τιμά η πρόσκληση συμμετοχή σε αυτήν εδώ την κοινοβουλευτική εβδομάδα. Και με χαρά μου εκπροσωπώ το Λετωνικό Κοινοβούλιο και θα σας μιλήσω για την εμπειρία που αποκομίσαμε στη Λετωνία από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η ιστορία της, η περίπτωση της Λετωνίας ήταν αντικείμενο και κριτικής και επένων τα τελευταία χρόνια και η ομιλία μου θα βασιστεί στα διδάγματα που αντλήσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ανάμεσα στο 2008 και το 2011 η Λετωνία έφτασε από μια κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ σε μια δυναμική εκπληκτική οικονομική ανάκαμψη. Το... Και για, τα... για να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά, η κυβέρνηση υιοθέτησε προγράμματα σε συνεργασία με τους διεθνείς δανειστές. Το πρόγραμμα, τα προγράμματα αυτά συνδέθηκαν με μη δημοφιλείς πολιτικές αποφάσεις και μέτρα λιτότητας και ως ε, αποτέλεσμα όμως των μέτρων αυτών οι κυβερνητικές δαπάνες εξισορροπήθηκαν με τα έσοδα και ξανακερδίσαμε την εμπιστοσύνη των διεθνών δανειστών μας. Είχαμε την ευκαιρία κατά τη διαχείριση της κρίσης να χρησιμοποιήσουμε δυνατότητες που μας έδιναν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Η Λετωνία κατά τη διάρκεια της κρίσης κατάφερε να χρησιμοποιήσει με καλύτερο τρόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι ώστε να τα διοχετεύσει στην, στο εργατικό της δυναμικό. Φυσικά όμως πάρα πολλά προβλήματα ανέκυψαν από τα μετραλιτότητα τα οποία επηρέασαν την οικονομική κατάσταση των επιμέρους ατόμων και της γενικής ε, ευημερίας. Σύμφωνα με δεδομένα από την Eurostat, ως αποτέλεσμα της ε, απότομης μείωσης των μισθών και των θέσεων εργασίας, το κατά μέσο όρο εισόδημα των ε, Λετωνών μειώθηκε κατά 28%. Και αυτό επηρέασε κυρίως δύο ομάδες, ε, τους νέους κάτω από 24 ετών και εκείνους από 45 έως 64 ετών. Για να μετριάσει αυτό να μετριαστούν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις, είχαμε μια στρατηγική, μια έκτακτη στρατηγική, το, ε, το κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας, το οποίο ήταν αποτελεσματικό στην ε, άμβλυνση των ε, κοινωνικών επιπτώσεων της ε, κρίσης. Είχαμε προγράμματα πρόνοιας για τις ε, οικογένειες, ιδίως τις οικογένειες με παιδιά. Επίσης, έγιναν πολλές δράσεις στις ε, αρχές της τοπικής ε, αυτοδιοίκησης και δόθηκε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση στους νέους. Και δόθηκε με αυτόν τον τρόπο και η δυνατότητα στους νέους και να διατηρήσουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να έχουν κάποιο εισόδημα. Ω αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, το κίνδυνος φτώχεια μειώθηκε κατά δύο φορές. Επίσης να πω ότι η στη Λετωνία παρουσιάστηκε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης για εργασία. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Λετωνών έφυγε στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης εργασίας. Στη Λετωνία το πρόγραμμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα θεωρείται ως ακρογωνιαίος λίθος. Το πρόγραμμα δηλαδή παλινόστησης των μεταναστών. Από το 2009 μέχρι το 2011 η ανεργία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ήταν σε απίστευτα υψηλά επίπεδα. Και τώρα το 35% των εργαζομένων κερδίζουν το βασικό μισθό και είναι στα όρια της φτώχειας. Αυτό μας δείχνει ότι η κρίση είχε πολύ βαριές επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό. Και το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι ένα καυτό πολιτικό θέμα. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, εφέτος εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μου για να μειώσουμε την ένδια των εργαζομένων και κυρίως μας ενδιαφέρει για αυτούς οι οποίοι έχουν οικογένεια και παιδιά και είμαστε έτοιμοι να μάθουμε και να αποκτήσουμε βέλτιστες πρακτικές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς φορείς όπως είναι ο ΟΣΑ. Γι' αυτό νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε ιδέες και προτάσεις για το πώς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην μείωση της ένδυας και να αντιμετωπίσουμε άλλα κοινωνικά προβλήματα στο σχέδιό μας κοινωνικής ανάπτυξης μέχρι το 2020 ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα επιτυχές πρόγραμμα μεταρρύθμισης και να βελτιώσουμε και την ευμάρεια των πολιτών μας. Είναι στόχος μας να μετακυλήσουμε το βάρος της φορολογίας από την εργασία σε άλλους συντελεστές. Επίσης θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την σκιώδη οικονομία Κάτι το οποίο βέβαια θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και είναι φανερό είναι φανερό ότι το θέμα της αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων θα παραμείνει ένα πάρα πολύ κεφαλαιόδες πρόβλημα και το 2013. Οι συστάσεις που έχουν διατυπωθεί δίνουν και την ανάγκη στην Λετωνία να πράξει περισσότερα για να μειώσει την ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να βοηθήσει την κοινωνική συμπερίληψη. Είναι πολύ σημαντικό για τα εθνικά κοινοβούλια να υποστηρίξουν όλες αυτές τις ενέργειες και να μπορέσουν να έχουν κάποια κοινωνική υποστήριξη και να εξασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση για τις ενέργειές του. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει σαν στόχο να βελτιώσει την συνέργεια μεταξύ ε, πολιτικής στα οικονομικά θέματα και στα θέματα απασχόλησης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να κατανοήσουμε ότι τα άτομα πρέπει να έχουν τον κεντρικό ρόλο. Θα πρέπει οι πολιτικοί να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η ένδια και η απασχόληση και η ανεργία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εξαρτάται πάντα από τι οικονομικέ συγκυρίες. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε μια αγορά εργασία με ενεργού συμμετέχοντε και να δώσουμε, δώσουμε κατά τις τομεί που έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν μελλοντικά απασχόληση σε πιο μόνιμο επίπεδο. Η συνεργασία με του κοινωνικού εταίρου λοιπόν θα μα βοηθήσει να έχουμε καλύτερα πρότυπα για την εργασία και όχι να οδηγηθούμε σε εργασία χαμηλή ποιότητα. οι εκθέσεις αξιολόγησης αντικτύπου γίνονται όλο και πιο σημαντικέ, ιδίω όταν ελείπουν οι απαραίτητοι πόροι. Έτσι, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι χρηματοδοτήσει στοχοθετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και κατά τη διάρκεια τη κρίση, αλλά και μετά την κρίση. Γιατί μετά από μια κρίση θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη και είναι απαραίτητο να αποφύγουμε υπερβολική αύξηση στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Τα συστήματά μας μετά από την κρίση είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Ήδη προχωρούμε σε μελέτες, κάποιες από τις οποίες χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα και θα χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα αυτών των μελετών για να καθαρίσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας. Έχουμε κάνει βελτιώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης στην ε, εκπόνηση πολιτικών και αυτό μας δίνει ελπίδα για το μέλλον με το να θεσπίσουμε πιο φιλόδοξους στόχους για τη βελτίωση της ευμάρειας των πολιτών μας. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν τα συμπεράσματα τα οποία έχουμε αποκομίσει από την κρίση. Θα πρέπει να υποφεληθούμε και από τις βέλτιστες εμπειρίες των άλλων χωρών. Δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε επί των επιτυχιών μας. Θα πρέπει να ε, προσελκύσουμε τους πολίτες που έφυγαν από τη Λετωνία να εξαγείρουν την πατρίδα τους και να έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ρεαλιστική μαρτυρία των εμπειριών σας από τη χώρα σας. Ε, θα ακούσουμε τώρα τον τελευταίο, την τελευταία βουλευτή, την Βερονίκα Φοντανιέ, που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχέση με την ετήσια ανασκόψη της ανάπτυξης για... Ευχαριστώ κυρία... Πράγματι την προηγούμενη εβδομάδα Νεκρίθη η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης με μια πολύ ευρία πλειοψηφία. Εμείς βασιζόμαστε σε 8 σημεία. Την ανάγκη να εγγυηθούμε την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση με διαφορετικές αλλαγέ και επενδύσει, τι λύσει για την ανεργία των νέων και είναι αυτό το οποίο μα απασχόλησε πάρα πολύ στο προηγούμενο πάνελ, μεταρρύθμιση των εργασιακών αγορών, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, την ανάγκη να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, να πετύχουμε το στόχο του να διατηρήσουμε δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας και να αντιμετωπίσουμε την ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όλα αυτά λοιπόν κατέληξαν σε μια συμβιβαστική λύση που μπορεί να μην ικανοποιήσει κανένα αλλά είναι αποδεκτή από όλους για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά θέματα στα πλαίσια της προσαρμογής. Τονίσαμε ιδιαίτερα τον κοινωνικό αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση σε βάθος σε σχέση με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής στα κράτη-μέλη που εξετάζει και τα αποτελέσματα και την, ε, την αξία τους. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν υποστηρίξει μια στεναρή εξυγίανση πέραν όλων των άλλων προβλημάτων και από την άλλη πλευρά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι ζήτησαν μια αύξηση των δαπανών χωρίς να σκεφτούν τα αποτελέσματα για την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Και υπάρχουν και φυσικά και ενδιάμεσες λύσεις και θέσεις και εκεί προσπαθήσαμε να εστιάσουμε περισσότερο αυτή την έκθεση. Η κρίση έχει υποχρεώσει τι χώρε μα να περάσουν σε πάρα πολύ σημαντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών του. Το 2009 και 2010 τα ελλείμματα τη ζώνη του ευρώ είχαν ξεπεράσει το 6% του ΕΠ και το δημόσιο χρέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είχε αυξηθεί από το 60% στο 90%. Εξάλλου, υπήρχε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, του κρατικού χρέους, που ξεκίνησε από τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών ορισμένων κρατών της ε, ζώνης του ευρώ και του κινδύνου να υπάρξει ρήξη τη ζώνη του ευρώ, όλα αυτά οδήγησαν στην ε, ανάληψη προγραμμάτων προσαρμογής που ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξα, αλλά είχαν πολύ επιθετικό χαρακτήρα και οδήγησαν σε μεγάλες θυσίες για τους πολίτες από τους οποίους πια δεν μπορούμε να ζητούμε περισσότερε θυσίε. Σε πολλα κρατήματα έχουμε φτάσει πια στο όριο αυτού που είναι ανεκτό από του πολίτε και έχουμε φτάσει στα όρια τη κοινωνική ανοχή η ανεργία στην Ευρωζώνη έχει φτάσει το 11,8% το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί άλλο, δεν μπορεί να είναι ανοιχτό και ορισμένε χώρε όπω δυστυχώ και η δική μου χώρα έχει φτάσει το 26%. Είναι ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση σε σχέση με του νέου. Όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, ο ένα στου πέντε νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργος ακριβέστερα το 22,8% και σε ορισμένα κράτη-μέλη ξεπερνάει το ποσοστό ανεργίας των νέων το 50%. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι αφόρητη. Η κατάσταση στον χώρο εργασία έχει επιδεινωθεί περαιτέρω το 2012 και η προβλέψει το 2013 δεν είναι αισιόδοξε. Έχει, έχει αυξηθεί ο κατακαιρματισμό τη αγορά εργασία η ανεργία μακράς διάρκειας έχει φτάσει ανησυχητικά επίπεδα, η, τα μέσα εισοδήματα των οικοκυριών μειώνονται σε πολλά κράτη-μέλη. Και επιπλέον οι δείκτες μας δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση να υπάρξει μεγαλύτερη και πιο βαθιά ένδυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένδυα και κοινωνικός αποκλεισμός, με μια αύξηση του ποσοστού των ενδεών μέσα στους εργαζόμενους και επίσης αυτό θα οδηγήσει σε μια βαθιά κοινωνική πόλωση στα κράτη-μέλη. Αυτή η κατάσταση που είναι δραματική και το γεγονός ότι σιγά σιγά αρχίζουν να διαλύονται οι για το ευρώ και το σενάριο της ε, κρίσης, η κατάσταση μάλλον για την κρίση του κρατικού χρέους είναι πιο ευνοϊκή από ό,τι πριν από μισό ή ένα χρόνο, χάρη και στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, όλα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στο να σκεφτούμε περισσότερο κατά πόσο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε τόσο αυστηρές προσπάθειες εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με λιγότερο επιθετικό τρόπο. Μέχρι τώρα έχουμε επιφέρει στον ασθενή μια θεραπεία σοκ, αλλά τώρα που είναι κάπως καλύτερα, ίσως είναι καιρός να αλλάξουμε τη θεραπεία και την ποσολογία. Στους επόμενους μήνες έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα προβλήματα γιατί οι οικονομίες μας έχουν ακόμα μεγάλη ε, μεγάλες αδυναμίες και ο κοινωνικός αντίκτυπος κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι προβλέψεις λένε ότι η Ευρώπη σιγά σιγά θα επανέλθει στην οικονομική ανάπτυξη μέσα στο 2013 και θα είναι πιο έντονη αυτή η ανάκαμψη μέσα στο 2014. Παρ' όλα αυτά, οι προβλέψεις αυτές δεν είναι ομοιόμορφες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο αντικές για τις χώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία του μνημονίου και ακριβώς είναι οι χώρες αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας και την επιδίδωση των κοινωνικών δικτών. Αυτές τις στιγμές που έχει βελτιωθεί η σταθερότητα στο χρηματοοικονομικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι που δεν πρέπει να τους παραγνωρίζουμε, η επιστροφή στον δρόμο της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητά μας. Είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και να αναθεωρήσουμε τις οικονομικές μας πολιτικές και είναι απαραίτητο να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της εξυγίανσης και της εδραίωσης των προϋπολογισμών και των οικονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τη κοινωνική πολιτική και των μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση από την άλλη πλευρά. Είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε λοιπόν τα προγράμματα εδραίωση των προπολογισμών για να μειωθούν τα ελλείμματα τα οποία παραμένουν ακόμα και για να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο χρέωση των κρατών μελών για να είναι και ε, βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά. Αυτό όμω πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι διαφοροποιημένο, θα είναι αναλογικό και θα ευνοήσει την ανάπτυξη. Αυτό ακριβώ δέχτηκε η Επιτροπή Απασχόλησης, ότι πρέπει να συνεχίσει η εξυγίανση των οικονομικών, αλλά να είναι διαφοροποιημένη, αναλογική με τι συνθήκε και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ανάκαμψη της οικονομίας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο ρυθμός λοιπόν της ε, εξυγίανσης και της προσαρμογή θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένος μεταξύ των χωρών επί τη βάση της δημοσιονομικής κατάστασης. Μια χώρα που έχει ένα χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ έχει πολύ περιορισμένο χώρο για να έχει ε, επεκτατικές πολιτικές προϋπολογισμού διότι είναι φανερό ότι η εξυπηρέτηση του χρέους δεν αφήνει αρκετό περιθώριο για κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, οι χώρε οι οποίε έχουν χαμηλό επίπεδο συνολικού χρέους μπορούν να εφαρμόσουν πιο εποφελώς τέτοια πολιτική, ιδίω σε εποχές κρίσης. Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει μία πανάκια, μία μοναδική συνταγή που μπορεί να ισχύσει για όλου. Δεν πρέπει επίση να ξεχάσουμε την ανάγκη να εξηγιάνουμε τα οικονομικά τα δημόσια, αλλά αυτή η διαδικασία εδραίωση στο επίπεδο του προπολογισμού δεν θα πρέπει να υποθηκεύσει τη δυνατότητα ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση στι χώρε μα. Δεν πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ένδια και κοινωνικό αποκλεισμό ή δεν πρέπει να υποσκάψει τι δημόσιε υπηρεσίε ποιότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τι χώρε οι οποίε βρίσκονται σε ύφεση ή δείχνουν δείκτε πολύ περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη και που έχουν ήδη κάνει πολύ σημαντικέ προσπάθειε για να βάλουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά του. Για τι χώρε αυτέ είναι πολύ σημαντικό, εάν είναι δυνατόν, να έχουν μεγαλύτερη ευκαμψία σε σχέση με τον ρυθμό που θα ακολουθηθεί για την προσαρμογή των δημοσιονομικών του. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Ολοκληρώνουμε έτσι τις διαφορές παρουσίες. Έχω αυτή τη στιγμή πέντε εγγεγραμμένους. Θα μας μείνει και κάποιος χρόνος, αν κάποιος άλλος ε, επιθυμεί να μιλήσει. Είστε ευπρόσδεκτοι, έχετε τη λευκή κόλλα μπροστά σας, μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο ή αλλιώς μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα η Βαρορίντε Κατάν, ο Κέθαν, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Απασχόλησης στη Βουλή των Λόρδων και που εδώ θα ανήκε στην ομάδα ECR των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστικών και μετά ο κύριος Πούπακης, Ευρωβουλευτής. Και Βαρώνη, κυρία Οκέθα, να έχετε το λόγο. Μάλιστα, να πω ότι καταθλίβομαι από την κατάσταση που μας παρουσίασαν στην Λετωνία είχαν πραγματικά προβλήματα και έκαναν πράγματα για αυτά, έλαβαν μέτρα. Και από ό,τι φαίνεται, κάθε κάτοικος της Λετωνίας ενδιαφέρθηκε για τη λύση και είμαι πολύ περίεργη να ακούσω περισσότερες πληροφορίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει το σκεπτικό οι νέοι που πηγαίνουν σχολείο με το Σάββατο να δουλεύουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κόσμο είχε πολλά χρήματα και δεν χρειαζόταν να εργαστεί για αυτά. Ο πρόεδρο τη αλυσίδα Τέσκο άρχισε δουλεύοντα ω μαθητή τα Σάββατα. Φορτώνοντα και ξεφορτώνοντα και φτιάχνοντα τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Και τώρα έχει γίνει ένα από του πιο σημαντικού και ισχυρού επιχειρηματίε στον κόσμο. Υπάρχουν μοντέλα τέτοια και έχουμε δει στο παρελθόν τέτοια παραδείγματα. Όμω είναι πολύ δύσκολο να δώσει κίνητρα στου νέου ανθρώπου να σηκωθούν νωρί το Σάββατο, να σηκωθούν από το κρεβάτι του και να πάνε για δουλειά. Είναι εύκολο ίσως σε μια μικρή κοινότητα όπως η δική μου να κάνεις κάτι τέτοιο, να δώσεις ένα κίνητρο σε ένα νέο και να του πει, εντάξει θα σου δώσω και αν έρθει να με βοηθήσει στις 10 το πρωί. Είναι πιο δύσκολο όμως σε μεγαλύτερες κοινότητες να δημιουργήσεις αυτήν την πειθαρχία στους νέους και να τους δώσεις αρκετά κίνητρα ώστε να το κάνουν αυτό. Και αναρωτιέμαι τι σκέφτονται και πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσφατα δημιουργήσαμε ένα νομοσχέδιο στο, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που έχει ψηφιστεί στο μεταξύ το οποίο θα ενθαρρύνει τις νεότερες γενιές να βρίσκουν απασχόληση στον τόπο διαμονή τους. Διότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πληθυσμό που γυράσκει πολύ γρήγορα. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μεγαλύτερη πειθαρχία στους ανέργους, να τους δώσουμε περισσότερες δεξιότητες, έτσι ώστε να τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στην αγορά εργασία. και εμεί ω η απερχόμενη γενιά εργαζομένων πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό. Ε, δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι θέλουμε να μας δώσει αυτά τα κονδύλια Ευρωπαϊκή Ένωση για να το κάνουμε αυτό ή θέλουμε να βοηθήσει η κυβέρνηση. Όχι. Από ό,τι μου λένε, κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούσε έναν επιπλέον Εάν κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση απασχολούσε έναν επιπλέον εργαζόμενο, δεν θα υπήρχε σχεδόν ανεργία. Γι' αυτό ας δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το διπλανό μας. Πώς μπορούμε να του απλώσουμε μια χείρα βοήθειας και να του πούμε πειθαρχή σου προσπάθησε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο συνάδελφος που, κύριος Πουπάκης ο οποίος είναι Έλληνα, ε, μέλο τη επιτροπή ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και μέλο του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εφαρμογή πολιτικών ακραία λιτότητα ω αντίδοτο στα κράτη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα αφενό δεν επέφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα όπω άλλωστε υπονόησε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την πρόσφατη παραδοχή του για λάθος συνταγή και αφετέρου αυτή η πολιτική υπονόμευσε την κοινωνική συνοχή δημιουργώντα μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ο μέχρι σήμερα απολογισμό των κοινωνικών επιπτώσεων στη χώρα μου την Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ένα στου τρει Έλληνε ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια, με το βασικό μισθό να είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια. Οι άστεγοι και τα σύντια πολλαπλασιάζονται. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 26% με ένα στου δύο νέου να βρίσκονται στο εργασιακό περιθώριο. Μία στι δύο οικογένειε αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι της, η φορολογία αυξάνεται, οι μισθοί μειώνονται και οι τιμές παραμένουν ίδιες ή και ανεβαίνουν. Δημοσιονομική λύση όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κοινωνική διάλυση, αφού οικονομία και κοινωνία είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Απαιτούνται λοιπόν κοινωνικά δίκαιες και αναπτυξιακές πολιτικές που θα ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και θα στηρίζουν σε κάθε περίπτωση τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση κατά το σχεδιασμό τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών στρατηγικών. Είναι φυσικά εκ των ουκάνευ ότι πρέπει να επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας μέσα στην Ένωση στη βάση της αλληλεγγύης, της στήριξης και συνεργασίας. Έχουμε ανάγκη τους εταίρους μας. Είναι χρέος όλων μας να διαφυλάξουμε τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ιδεώδη, δίδοντας ελπίδα και προοπτική σε όλους ανεξαιρέτως τους Ευρωπαίους Συμπολίτε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο συναδελφός μας Ζωζέ Βιραντασίλβα, πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Προσαρμογής στην Πορτογαλία και μέλος του Σοσιαλιστών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την συμπέληψη αυτού του σημείου στην ημερησία διαταξή μας και θα ήθελα με απλό τρόπο, απλοποιημένο τρόπο να εντοπίσω τις, τα τρία κύρια επίπεδα επίπτωσης της διαδικασίας δημοσιονομικής προοπτικής προσαρμογής μάλλον, που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία, όπως και πολλές άλλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συνοπτικά, η πρώτη πτυχή είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του απογεύματος, το ότι δεν είναι σε θέση η αγορά εργασίας να προχωρήσει στην ανανέωση των γενναίων. Λέμε στην όπως είπαμε σήμερα, στην Πορτογαλία, όπως και σε άλλες χώρες, είναι κλειστή η αγορά εργασίας για τους νέους. Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού ε, ανέργων μεγάλη ηλικία οι περισσότεροι που βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση που είναι πολύ νέοι για να συνταξιοδοτηθούν, αλλά και πολύ ηλικιωμένοι για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα <clears throat> το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται. Ένα τρίτο θέμα είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την <clears throat> σταθερή διάβρωση των ελάχιστων κοινωνικών επιπέδων που είναι αποτέλεσμα των μνημονίων και των συνταγών που συζητήθηκαν και έτυχαν διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φορέων που τους δίνουν χρηματοδότηση. Θα ήθελα να σταθώ για κάθε ένα από αυτά τα τρία προβλήματα με λίγα λόγια. Η ανεργία των νέων, η ανεργία των πιο ηλικιωμένων και η υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων. Θα σας διαβάσω ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την απασχόληση των νέων έλεγε το κείμενο αυτό, το οποίο μετά θα σας πω από ποια χρονική εποχή προέρχεται. Το να δώσουμε μια νέα ευκαιρία σε όλους τους νέους πριν καλύψουν 16 μήνες ανεργίας με τη μορφή της κατάρτισης, της ε, ε ανακύκλωσης ή της παροχής ε, ε, δυνατοτήτων εργασίας και μαθητείας για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας. Αυτή ήταν η πρώτη κατευθυντή γραμμή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το 1997. Χρησιμοποιήθηκε για τα επόμενα χρόνια στα σχέδια απασχόλησης. Κάποια στιγμή μειώθηκε στους τέσσερις μήνες αυτό το χρονικό διάστημα και υπήρξε μια κοινή δέσμευση που είχε αναλυθεί από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια χρονική στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί αυτή τη νέα σύσταση για την αγίηση για τους νέους που ήταν πολύ κοντά σε αυτή την ε, κατευθυντήρια γραμμή του 1997 ίσως θα πρέπει να αποδειθούμε όλοι σε κάποια περισσότερη σκέψη για το τι έγινε στην Ευρώπη ώστε αυτή η στρατηγική η οποία ήδη είχε αν είχε αντιμετωπιστεί το 1997, δεν είχε καμία επιτυχία. Δεν πρόκειται εδώ να οικοτολογήσω για το θέμα αυτό, γιατί δεν έχω και χρόνο, αλλά νομίζω ότι τα τρία βασικά θέματα εδώ ήταν η μείωση της πολιτικής σημασίας καταρχήν του προβλήματος αυτού. Το γεγονός επίσης ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και τρίτον, το γεγονός ότι υπήρξαν άλλες πραγματικότητες οι οποίες σε ό,τι αφορά την επεξεργασία της ευρωπαϊκής πολιτικής έχουν καταλάβει το χώρο που είχε παλιά η κοινωνική πολιτική. Με τον τρόπο αυτό τα κοινωνικά θέματα έχουν υποβαθμιστεί σε σημασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμα σε ό,τι αφορά τα θέματα των ελαχίστων κοινωνικών προτύπων. Αναφέρθηκε ήδη το πρωί ότι 19 από 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια έχουν δει να αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών τους που βρίσκονται σε κατάσταση ένδυση. Ακόμα πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι 11 από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαν να μειώνεται το κατόφλι της ένδυας. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια μεγάλη ομάδα από χώρε μείωσε την ονομαστική αξία σε τρέχουσες τιμές του κατοφλίου της ένδυας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι πολύ δύσκολο ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα στους νέους όταν υπάρχει τόσο μεγάλο τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων σε ανεργία και όταν αυξάνεται συνέχεια η, ανεργία, η, ένδια σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάλι ο κύριος Αλεξάνδρας Σέρκας. έχει ήδη μιλήσει, είναι μέλος των Ισπανών Σοσιαλιστών. Έχω ήδη κάνει κάποια σχόλια κυρία Πρόεδρε στην προηγούμενη σειρά παρεμβάσεων και ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τότε την ανεργία μου για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε να εξελίσσονται τα στοιχεία στις χώρες αυτές που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, πως καταργούνται και καταστρέφονται όχι μονάχα τα ατομικά δικαιώματα αλλά και τα συλλογικά δικαιώματα. Θέλω να κάνω τώρα δύο πάλι παρατηρήσει. Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξή. Οποιοδήποτε έμφρον άτομο γνωρίζει ότι μια πολιτική θα πρέπει να εκτιμάται και να κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα και όχι μονάχα τις προθέσεις. Αν η πολιτική η οποία εφαρμόζεται στις χώρες μας μετά από τέσσερα χρόνια κρίσης μας δίνει περισσότερη ε, ανεργία, περισσότερες μακροοικονομικές ε, ανισότητες, περισσότερες κοινωνικές ανισότητες και μεγαλύτερη ένδια, όπως αναφέρθηκε από όλους. Αυτά, λοιπόν, δεν μας δίνουν περιθώριο παρά να συμπεράνουμε ότι είναι μια λαθασμένη πολιτική. Αυτό είναι θέμα πραγματικών στοιχείων, δεν είναι θέμα ιδεολογικής προσέγγισης. Οι γνώμες είναι κάτι το οποίο είναι στην κρίση του καθενός. Αλλά τα δεδομένα μας αντιμετωπίζουν κατά πρόσωπο με μια δραματική πραγματικότητα που μας λένε ότι ξεκινώντας με τη λιτότητα του προϋπολογισμού, ξεκινώντας από την ε, περισταλτική αντιμετώπιση των δημοσίων δαπανών, υποτίθεται ότι με όλα αυτά θα αυξανόταν η απασχόληση, η, θα, ήταν, θα προέκυπτε ανάπτυξη, νέες πιστώσεις κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι πριν από 4-5 χρόνια, πίστεψα καλή την πίστη ότι θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλοί πιστέψανε, ανεξάρτητα από πολιτική παράταξη, ότι ο ορθολογισμό τη αγορά θα οδηγούσε σε κάποια θετικά αποτελέσματα. Αλλά είναι γεγονό ότι δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Χθε ο Επίτροπο Όλη Ρεν μίλησε για μια ευελικτοποίηση, να γίνει πιο ευέλικτο ο μηχανισμό προσαρμογή και ο ρυθμό τη προσαρμογή. Γιατί η ακαμψία που ακολουθήθηκε έχει οδηγήσει σε μαθηματική καταστροφή χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Δεν υπήρχαν χρήματα παρά μόνο για να πληρώνουν το δημόσιο χρέος. Το γεγονός ότι τα spreads σε ορισμένες χώρες αυξήθηκαν αστρονομικά, αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε καταστροφικό αποτέλεσμα. Το κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές στην Ισπανία θεωρούσε ότι αν έρθει στην εξουσία και εφαρμόσει σωστά αυτή την πολιτική προσαρμογή, οι αγορέ θα συμμορφωνόντουσαν και θα δίναν την εμπιστοσύνη σου. Αυτό δεν έγινε. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει είναι διπλάσια από ό,τι όταν ήρθε στην εξουσία η κυβέρνηση Ραχώη. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθήθηκε. Κάτι έλειψε, κάτι πήγε στραβά. Γιατί δεν έχουμε τώρα το ηθικό ανάστημα να καταλάβουμε και να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Είναι απόλυτα σαφές ότι έχουμε κάνει κάτι ότι έχουμε κάνει ένα τέτοιο μεγάλο λάθος. Είναι τρομερό στη χώρα μου ότι δεν υπάρχουν καθόλου χρηματοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να πληρώνουν με επιτόκια δυο και τρεις φορές πιο ψηλά από αυτά των γερμανικών εταιριών. Όταν έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Γιατί η ορθόδοξη αυτή αντιμετώπιση του μνημονέου έχει στερέψει κάθε, κάθε πίστοση ο κόσμος πέφτει σε απόλυτη αδράνεια γιατί δεν υπάρχει εσωτερική ζήτηση. Ο κόσμος έχει μια κοινή λογική, όμως καταλαβαίνει ότι αυτά δεν πάνε πουθενά. Γι' αυτό, εάν δούμε λιγάκι πιο κριτικά, με κριτικό πνεύμα, αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε τα τέσσερα χρόνια που περάσανε, είναι απαραίτητη. Δεν λέω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική προσαρμογής. Είχαμε 60% του ΑΕΠ χρέο όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και τώρα έχουμε 100%. Υπάρχει αυτή η πολιτική η οποία οδήγησε και η οποία εμπόδισε την εσωτερική ζήτηση και την κατανόηση στη χώρα μας. Κλείνουν οι επιχειρήσεις και κάθε φορά ρίχνουν ε, χιλιάδες άνεργους στην, ε, στον δρόμο. Τρεις χιλιάδες κάθε μήνα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 55% νέων που είναι άνεργοι και ένα πολύ ψηλό επίπεδο γενική ανεργία. Όλα αυτά έχουν τεράστιε συνέπειε, όχι μόνο την απασχόληση, αλλά και στο υγειονομικό σύστημα, στο σύστημα. Το Ο κόσμο δεν μπορεί να αγοράσει φάρμακα πια. Χάνουν τα δικαιώματά του, χάνουν τη δυνατότητα να αγοράζουν τα βασικά αγαθά. Αλλά κυρίω το βασικό είναι ότι καταστρέφεται ο κοινωνικό σύστημα, ο κόσμο χάνει την εμπιστοσύνη του και την ελπίδα. Δεν είναι ένας αλγόριθμος μονάχα η οικονομία. Είναι και η εμπιστοσύνη του κόσμου στην ε, κοινωνία και στη δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί, έχει καταβαραθρωθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην Ευρώπη. Λοιπόν, πέρα από κάθε ιδεολογία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτι δεν λειτουργήσε καλά. Ότι έλειψαν πράγματα από αυτή την πολιτική προσαρμογής διότι έχουμε καταλήξει σε μια κατάσταση απόλυτα δραματική σε πολλές χώρες. Και την πληρώνουν την ύφη αυτοί που δεν έχουν καμία ευθύνη για την κρίση. Ενώ το City του Λονδίνου, η Wall Street και όλοι αυτοί, αυτοί δεν πάθανε τίποτα, έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα τρία χρόνια για να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την δική τους κερδοφορία και τα στοιχεία της κρίσης που οφείλεται καθαρά στις δικές τους ενέργειες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας άφησα να μιλήσετε περισσότερο, θα παρατηρήσετε επειδή έχουμε χρόνο. Καλό τους τελευταίους που δεν έχουν γραφεί ακόμα και που θα επιθυμούσαν να μιλήσουν να μας κάνουν σήμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Διαφορετικά θα δώσω το λόγο στην Ένε Τσούμπερ ως τελευταία ομιλήτρια αυτού του πάνελ. Είστε ευρωβουλευτής από την ομάδα της Γκουε και έρχεστε από την Πορτογαλία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ε, κρίση και τις επιπτώσεις στον τομέα της ε, απασχόλησης. <clears throat> Αναφέρονται όλα αυτά στην έκθεση της Κομισιόν και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι κάποιες από τις συστάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν στο εγγραφό αυτό δεν έχουν βελτιώσει, έχουν μάλλον επιδεινώσει την κατάσταση εργασίας στις χώρες οι οποίες είναι πιο αδύνατες οικονομικά, κυρίως στις χώρες του μνημονίου. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Η ευκαμπτοποίηση των συνδικών εργασίας οδήγησε στην επισφαλή εργασία που οδηγεί μαθηματικά και στην ανεργία. Η μείωση των αποζημιώσεων απόλυσης θεωρήθηκε ότι ήταν ένας τρόπος δημιουργίας απασχόλησης. Αλλά οδήγησαν σε περισσότερες απολύσεις. Ο καθορισμός των αποδοχών σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε μία μείωση των ε, μισθών και ουσιαστικά φέρνει στους ώμους των ε, εργαζομένων την ευθύνη για την αύξηση της παραγωγικότητας που ξέρουμε ότι δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν επίπτωση στο θέμα αυτό. Αλλά επειδή μειώνονται οι αποδοχέ των εργαζομένων, όλα αυτά μειώνουν και το, την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού και επομένω αυτό οδηγεί όλη την οικονομία σε μία ύφεση. Στη χώρα μου λοιπόν, στην Πορτογαλία, προέβλεπαν οι συστάσεις του προηγούμενου εξαμείνουν να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Υπάρχουν τρει-τέσσερι τρόποι να το κάνει αυτό. Ή θα μειώσει κανεί τα κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα, ή θα μειώσει τι αποδοχέ, ή θα απολύει κόσμο. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για το κοινωνικό αντίκτυπο εδώ των πολιτικών που ακολουθούνται για την εξυγίανση των οικονομικών και τα μέτρα των μέτρων λιτότητος. Αλλά υπάρχει και μία άλλη όψη αυτών των μέτρων που είναι η δημιουργία κοινωνικών ε, ανισοτήτων και η όξυνση των ανισοτήτων. Στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, μειώθηκε το, το μερίδιο των ε, εισοδημάτων από μισθωτή εργασία σε επίπεδο, στα επίπεδα του 1984. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η πρόσοδος από την οικονομία πηγαίνει σε άλλους και όχι τους εργαζομένους. Συγχρόνως έχουν αυξηθεί η, τα κέρδη των επιχειρήσεων, έχει αυξηθεί το επίπεδο κερδοφορίας ορισμένων και, κέριων τομέων όπως είναι η τηλεπικοινωνίες, οι, εταιρείε οι εταιρείες ηλεκτρικής ε, παραγωγής και διανομής, όλα αυτά δείχνουν να υπάρχει μια δυτή κατά κάποιο τρόπο κοινωνία. Από τη μια μεριά μειώνεται η δυνατότητα, η αγοραστική δύναμη των ε, εργαζομένων και το εισόδημά τους, από την άλλη πλευρά αυξάνονται τα κέρδη ορισμένων επιχειρήσεων. Όλα αυτά μας κάνουν να βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστικά μια μεταφορά περιουσίας από τους εργαζόμενους στον κόσμο του κεφαλαίου. Κάτι ακόμα για αυτή τη συζήτηση. Μου φαίνεται εντυπωσιακό το ότι εξακολουθούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται καταστρέφουν κάθε μέρα θέσεις εργασίας. Κάθε μέρα καταστρέφονται 300 θέσεις εργασίας στην Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανάπτυξη τη στιγμή που ούτε καν βρισκόμαστε σε στασιμότητα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξαναγυρίσουμε σε ένα ευνοϊκό κλίμα για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη αν συνεχίσουμε με αυτές τις συνθήκες στον τομέα της αγοράς. Και ένα από τα θέματα τα οποία για μένα είναι θεμελιώδες, όταν μιλάμε για, για οικονομική ανάπτυξη, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς δημόσιες επενδύσεις, γιατί χωρίς δημόσιες επενδύσεις δεν θα επενδύσει και ο ιδιωτικός τομέας και με την πίεση που βρίσκεται στον κρατικό προπολογισμό δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δημόσιε επενδύσει. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά και έχουμε τονίσει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δημόσια επένδυση για να υπάρξει ανάκαμψη. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω λοιπόν είναι ότι πέρα από τα λόγια μας είναι απαραίτητο να αναστρέψουμε την κατεύθυνση των πολιτικών που ακολουθούμε. Πίσω από αυτά τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε όλοι υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι, ζωές κατεστραμμένες που δεν μπορούμε να τις παραγνωρίσουμε. Μία πολιτική η οποία θα αυξήσει την δυνατότητα, την ε, κατανάλωση και θα δώσει δυναμικότητα στην οικονομία είναι το να υπάρξουν περισσότερες δαπάνες σε τομείς κοινοφολιούς χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να δίνουμε κέρδη στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε κλειδωμένοι μέσα σε μια ιδεολογική προσέγγιση η οποία δεν οδηγεί σε τίποτα παρά μόνο σε περισσότερα κέρδη από την πλευρά των ε, ιδιωτικών εταιριών και του κεφαλαίου. σε βάρος του ίδιου του κράτους και σε βάρος των πολιτών, το οποίο καλείται πάντα να πληρώνει την ύφη στο τέλος. Και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει κανείς αντιμετωπίσει. Γιατί οι χώρες αυτές έχουν αφαιρέσει το εισόδημα των εργαζομένων στο όνομα του να καταβάλουν το χρέος τους, να πληρώσουν το χρέος τους, ενώ το χρέος αυτό συνεχίζει να αυξάνεται στις χώρες αυτές. είναι όλο και πιο δύσκολο το κρατικό χρέος για να το αποπληρώσει κανείς και δεν γίνεται καμιά προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθηκαν εδώ. Νομίζω ότι ο λαός της Πορτογαλίας και οι εργαζόμενοι των χωρών που βρίσκονται στη, στα μνημόνια αξίζουν μια μεγαλύτερη αναγνώριση γιατί αγωνίζονται και συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της, ε, των υπερβολικών κερδών και της διάβασης των δικαιωμάτων τους. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε στο σημείο που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ονομάζουμε Catch the Eye. Σημαίνει ότι όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να σηκώσει το χέρι του για να μιλήσει. Αν κάποιος από εσά θα ήθελε να μιλήσει, να αλληλεπιδράσει, να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν, Διαφορετικά θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες βουλευτές μας. Αυτός ο τίτλος σας δόθηκε, θα το κάνουμε με αντίστροφη σειρά σε σχέση με το τι κάναμε στην έναρξη τη συνόδου μας. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Φωντάνια και μετά στον κύριο ε, στην κυρία Ζερά. Μην αλλάξετε θέσεις. Βερόνικα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν πρέπει να είμαστε και τόσο απεσιόδοξοι όπως ο αγαπητός μου Αλέξανδρος Φέρκας. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε λιγάκι καλύτερα και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε και φυσικά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν είναι θετικά. Δεν πρόκειται τώρα να επανέλθω σε όλα αυτά τα οποία είπαμε ότι είναι απαραίτητη η εδραίωση του προπολογισμού, αλλά πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο χαρακτήρα. Σε αυτό το θέμα όλοι συμφωνούμε αυτή τη στιγμή. Επίσης όμως θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα πνεύμα εμπιστοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι εάν αποκτήσουν την εμπιστοσύνη θα αλλάξει η δυναμική. Και θέλω να απαντήσω τώρα στην Βαρονέσα η οποία μιλούσε για την πειθαρχία εργασίας των νέων. Οι νέοι μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τι είναι η πειθαρχία της εργασίας, αν έχουν εργασία και αν τους δώσει κανείς τις απαραίτητες πληροφορίες. Στη δική μου χώρα υπάρχει μια ένωση σε επίπεδο γειτονιά, η οποία εργάζεται μαζί με τους νέους, με νέους που είναι ανάπηροι, με νέους που έχουν προβλήματα ενσωμάτωση σε κοινωνικό επίπεδο. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν αυτό το υπόδειγμα συνεργασίας, έχουν κάνει πολλά εργαστήρια για καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση και μπορούν με τον τρόπο αυτό να έχουν και κάποια ε, χρηματοδότηση κάποια, κάποιες αποδοχές. Υπήρχαν πολλοί νέοι οι οποίοι ήταν ανάπηροι και δεν είχαν απολύτω τίποτα να κάνουν όλη μέρα και σηκωνόταν δύο η ώρα το απόγευμα. Από τότε που εργάζονται σε αυτά τα εργαστήρια είναι ήδη από το πρωί και θέλουν να μπουν μέσα και να εργάζονται. Γιατί έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον τους και έχουν ελπίδες. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε την ελπίδα αυτή στους νέους. Είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με τα διορθωτικά ταμεία την ε, υποστήριξη αυτών των πρωτοβουλειών που γίνονται σε κράτη-μέλη όπως η δική, η δική μου χώρα που δεν μπορούν από μόνα τους τα κράτη αυτά να λύσουν τα προβλήματα αυτά και δεν βλέπω να υπάρχει καλύτερη χρήση των ταμείων αυτών και των κονδυλίων παρά μόνο για να βοηθήσουν να δουλεύουν οι νέοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο τον Βίλα ε, Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση όμως πριν δώσω το λόγο γιατί αναφέρθηκαν δύο κατά την άποψή μου πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον το για την αποκατάσταση της κατάστασης πόσο δύσκολο πόσο σημαντικό ήταν η μόκλευση που προσέφερα τα διερθρωτικά ταμεία στη χώρα σας και πόσο αυτό συνδέεται με τις δημοσιονομικές προοπτικές θα δεσμευτεί το 25% της πολιτικής συνοχής υπέρ του, ταμείου, του κοινωνικού ταμείου. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης. Πάντα μου έκανε εντύπωση όταν ήμουν νέα είχα μάθει ότι ο Λένιν έλεγε ότι όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους ψηφίζουν με τα πόδια τους. Και όταν λέτε ότι το 10% των κατοίκων της Λιθουανίας ε, εγκατέλειψαν τη χώρα τους και δυσκολεύεται τόσο πολύ να τους κάνετε να επιστρέψουν. Πώς αμφισβητείτε τη συνταγή που εφαρμοστήκε στη χώρα σας. Θεωρείτε... Ξέρετε, η χώρα σας πάντα θεωρείται παράδειγμα. Κοιτάξτε, λέμε πάντα... Ε, η υπέστη λιτότητα, η ανεργία μειώθηκε, αλλά το τίμημα για αυτό ήταν τεράστιο. Όχι μόνο 10% των κατοίκων εγκατέλειψαν τη χώρα, αλλά μεταξύ αυτών σίγουρα και πολλοί νέοι. Θεωρείτε ότι αυτή ήταν η σωστή τακτική. Πώς θεωρείτε ότι σχετίστηκε το κοινοβούλιο της χώρας σας με την επεξεργασία αυτής της συνταγής του, του μνημονίου που εφαρμόσε το Λετωνικό Κοινοβούλιο που χρειάστηκε να εφαρμόσετε στις διάφορες νομοθεσίες. Για να το πω πιο σαφώς, θεωρείτε ότι το Λετωνικό Κοινοβούλιο ε, έδωσε επαρκώς τη γνώμη του όταν εφαρμόστηκε η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολλέ ερωτήσει με κοβλήθηκαν. Όσον αφορά την επιστροφή της Λετωνίας στο δίλημα ανάμεσα αξιολόγηση ή κρίση. Ε, να πω ότι η κυβέρνησή μας επέλεξε τη σωστή πορεία, την πορεία της αξιολόγησης. Το μόνο που ίσως κάναμε με διαφορετικό τρόπο θα ήταν να μην επιτρέπαμε στους ε, λετονούς να δανείζονται τόσο πολύ χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες. Αυτός ο υπέρμετρος δανεισμό ήταν και ένα από του λόγου τη κρίση. Ο κόσμο δεν μπορούσε να πληρώσει το δανειό του. Όντω τώρα σε αυτό που είπατε το 10% είναι ένα τίμημα που πληρώσαμε. Απόλυας πληθυσμού και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέχρι 35 ετών. Οι άνθρωποι δηλαδή που ήξεραν ότι υπάρχουν ευκαιρίες έξω από τη Λετωνία και που δεν είχαν έτσι κι αλλιώς δυνατότητες στη Λετωνία να βρουν δουλειά. Το σχέδιο ανάπτυξης λοιπόν για τη Λετωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση είναι ελπιδοφόρος σχετικά. Αν δείτε κιόλας ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες γίνονται περικοπές μισθών, τα τελευταία χρόνια οι μισθοί αυξήθηκαν στη Λετωνία. Και συνεχίζεται και φέτος αυτή η αύξηση στους μισθούς. Και σε άλλες χώρες λοιπόν θα ήθελα να υπήρχαν τέτοια μέτρα εξυγίανσης Φυσικά και χρειάζεται να υποφέρεις, αλλά από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει ανάκαμψη, όπως στη Λετωνία και ότι πολλές εταιρείε προχωρούν στην εξυγίανση των οικονομικών τους, αυξάνουν τους μισθούς και αρχίζουν να επιστρέφουν οι μετανάστες ιδιαίτερα για να εργαστούν σε εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό τομέα, σου δίνει δυσεδοξία. Επίσης, στη Λετωνία έγινε ολική αναδιάρθρωση της οικονομίας μας. Οι εξαγωγές μας ήταν ε, το 20% του ΑΕΠ πριν την κρίση. Τώρα οι εξαγωγές μας αποτελούν το 80% του ΑΕΠ. Έχει γίνει λοιπόν πολύ ανταγωνιστική η Λετωνία. Τώρα όσον αφορά τα ταμεία που αναφέρατε και την ε, κατανομή των κονδυλίων στο μέλλον, να σας πω ότι για τη Λετωνία όλα τα ταμεία είναι σημαντικά. Το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο για τη Γεωργία, παρότι λαμβάνουμε λιγότερα κονδύλια από τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μία έκκληση θα ήθελα να κάνω στην Επιτροπή. Μην κάνετε περικοπές στο Ταμείο για τις Επιστήμες. Είναι η μόνη ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας μας και ανάκαμψη. Είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα αυτών που θα δώσουν προστιθέμενη αξία και σε αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάζουμε να πάμε την ανακαμψή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, εξωτιμε κύριε. Αυτή είναι η φιλοδοξία της χώρας σας. Σας ευχόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Τελευταίος εμπειρογνωμών βουλευτής, ο Ζωζέ Μανώλη Καρναβάρο, της Επιτροπής ε, Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης του Κοινοβουλίου. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η κυρία Φοντέν Λοπέ. Σίγουρα είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα απορίσματα αυτών των μελετών. Με τον τρόπο αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και κάποια, κάποιο συνδυασμός της εργασίας με τις ακαδημαϊκές με τις ε, ακαδημαϊκές σπουδές. που φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό μετά από μια ορισμένη ηλικία να μπορούν τα άτομα να συνδυάζουν ε, ακαδημαϊκή εμπειρία με επαγγελματική ε, εμπειρία. Όλα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν μια κατάλληλη εργασία. Φαίνεται εδώ πέρα από τη συζήτηση το γεγονό ότι οι περισσότερε παρεμβάσει, τα 85% των παρεμβάσεων ήταν από εκπροσώπου των χωρών του Νότου, δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα από τη διαδικασία προσαρμογή και λιτότητα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Ντασίλβα, παρά το γεγονό ότι δεν προέρχεται από την ίδια παράταξη όπω εγώ, ότι συμφωνώ ότι υπήρξαν πραγματικά σημαντικές επιπτώσεις από τις ε, ενέργειες προσαρμογής και αυτό οδήγησε σε δυσκολία πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς μια θέση εργασίας και ιδίως για αυτούς που είναι κοντά στην σύνταξη και υπήρξαν και κάποια, κάποιες υποβαθμίσεις στα επίπεδα των, ε, των δικαιωμάτων. Έχουμε μια διάγνωση λοιπόν η οποία δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να διαφυσβητήσω και φυσικά η πορτογαλική κυβέρνηση έκανε μέτρα για να την αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Με την κυρία Ζούμπερ τώρα βέβαια υπάρχουν επί της ουσίας κάποια πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση του χώρου εργασίας και θα οδηγούσε σε πρώτη φάση σε μια μείωση της απασχόλησης. Η πορτογαλική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η αύξηση της ανεργίας ξεπέρασε λιγάκι αυτά τα οποία προβλεπόταν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο δρόμος αυτός είναι ο σωστός. Και δεν συμφωνώ με αυτά που έλεγε για τις επενδύσεις, ότι πρέπει να γίνουν όλα με δημόσιες επενδύσεις. Πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα πρέπει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα κοινωτικά κονδύλια και επίσης να προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό της Πορτογαλίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα οι επενδύσεις από το εξωτερικό και προφανώς αυτές οι επενδύσεις λόγω της κρίσης δεν μπόρεσαν να φέρουν πόρους αλλά θα πρέπει να ψάξουμε και άλλες από τις παραδοσιακές πηγές επενδύσεων για την Πορτογαλία. Επίσης και με τον κύριο Σέρκας, εγώ δεν είμαι τόσο ε, απεσιόδοξος. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια μεγαλύτερη ευκαμψία στους μηχανισμούς προσαρμογής. Αυτό ισχύει και για την Ισπανία και για την Πορτογαλία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιβυρική αλληλεγγύη για τα θέματα αυτά. Δεν είναι μονάχα για γεωγραφικού λόγου, αλλά επειδή είναι παρόμοιε σε μεγάλο βαθμό οι καταστάσει τη χώρα μα και οι διαδικασίε. Για τον κύριο Πουπάκη. Κατανοούμε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερε οι δυσκολίε από ό,τι στην Πορτογαλία και την Ισπανία και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μας με την Ελλάδα, όλα αυτά μπορούν να επιληθούν μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μεγαλύτερη συνεργασία που είναι ζωτικού χαρακτήρα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Η Πορτογαλία είναι ακόμα μια κατάσταση η οποία είναι εν εξελίξη, δεν έχουν κλείσει τα θέματα αυτά, αλλά όλα αυτά που αναφέρθηκαν από τον γείτονά μου εδώ στα αριστερά είναι λύσεις που προσπάθησε να εφαρμόσει και η Πορτογαλία. Κάθε λαός βέβαια έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τις ιδιοσυγκρασίες του. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρει κανείς απόλυτα αυτά τα οποία έχουν λειτουργήσει σε μια χώρα σε μια άλλη χώρα. Κάναμε και τις δικές μας, είχαμε και εμείς τις εμπειρίες μας σε σχέση με τη λιτότητα και την μείωση του δημοσίου ε, ελλείμματος. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν και σε ε, συμφωνία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός λαού και συγχρόνω μέσα στο πλαίσιο τη Ευρώπη, γιατί η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Euh. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και στις δύο αυτές συνόδους. Για αυτή τη δεύτερη σύνοδο θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα Συμφωνώ με τους προβληματισμούς του συναδελφού Καναβάρου. Στον πρώτο γύρο τραπέζης ε, είχαμε μια γεωγραφική ισορροπία όσον αφορά τις παρεμβάσεις και ενώ στη δεύτερη σύνοδο επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε χώρες όπου το ζήτημα της απασχόλησης αποτελεί εθνικό πρόβλημα και φυσικά άκουσαν και οι υπόλοιποι μέσω της συζήτησης ε, αυτό ήταν ούτω ή άλλω ο σκοπό μια τέτοια συνόδου. Θα ήθελα να κάνω πέντε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, πέρα των όσων λένε σήμερα οι εμπειρογνώμονε για το πολλαπλασιαστική επίδραση, ο τρόπος επεξεργασίας των προγραμμάτων προσαρμογή στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι αφετέρου, καθώς και οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβούλων, όλοι αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, διαδικασίας επεξεργασίας, όλα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή των μεταρρυθμίσεων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δεδομένων όλων αυτών δεν ξέρουμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Διότι φυσικά στις χώρες όπου σήμερα η κρίση έχει καθιερωθεί με τρόπο μετακίνητο είναι οι χώρες χώρες όπου είναι πιο περίπλοκη η συνεργασία, η συλλογική επεξεργασία από τις χώρες που αντιμετωπίζουν λιγότερο κρίσιμα προβλήματα. Δεύτερη παρατήρηση στην αρχή της κρίσης, ΜΑΜΑ μεταξύ του 2007 και του 2008, ότι εμείς εδώ, σε Ευρωπαίοι, λέγαμε «Α, είναι αμερικανική η κρίση» και εν τέλει στην Ευρώπη δεν έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες. Μεταξύ άλλων, διότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές μας θα μας επιτρέψουν να αποσβέσουμε την κρίση. Αυτοί οι αυτόματοι σταθεροποιητέ, ε, μη βάρβαρο, η ορολογία σημαίνει αυτό το σύστημα κοινωνική προστασία. Και αυτό που κάνει εντύπωση ότι μόλις 4 5 χρόνια αργότερα ξεχάσαμε αυτά που λέγαμε τότε, τότε που ξεκίνησε η κρίση. Διότι κοιτώντα τα προγράμματα προσαρμογής που ακριβω πολύ συχνά επηρεάζουν πρώτα απ' όλα αυτού τους αυτόματου σταθεροποιητέ, όπου έπρεπε πρώτα απ' όλα να αναρωτηθούμε πώς θα επινοήσουμε νέους σταθεροποιητές αυτόματους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι κάτι ξεχάσαμε. Με άλλα λόγια, σκεφτήκαμε τόσο βραχυπρόθεσμα που δεν λάβαμε αρκετά σοβαρά τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις. Και αυτό ανακαλύπτουμε ξαφνικά τώρα, σε αυτό βρισκόμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή, όταν συζητάμε πολλαπλασιαστές. Η τρίτη μου παρατήρηση είναι ότι θα ήθελα να πω στους ε, εκπροσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ήδη πολλές φορές ε, ζητάμε όταν υπάρχει μια τρόικα η οποία παρεμβαίνει σε ένα κράτος μέλος αυτή η τρόικα να μετατρέπεται σε κουαρτέτο να συμπεριλαμβάνει δηλαδή εκπροσώπους ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου Πολλές φορές έχουμε συναντηθεί με αυτόν τον οργανισμό, το Διεθνή Οργανισμό εμπόριο. και εκεί υπάρχουν ομάδες ε, έτοιμοι, εμπειρογνώμονες να παίξουν στο κοινωνικό τομέα το ρόλο που παίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλής η θέση αυτή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αξίζει την υποστήριξή μας και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε ενδεχομένως να έχουμε μια πιο καθολική προσέγγιση των ε, προγραμμάτων προσαρμογής. Η τέταρτη μου παρατηρήση αφορά ε, τα όσα λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο συμβουλίου. Ακούστε τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το απόγευμα όσον αφορά το Συμβούλιο ε, υποθέσεων απασχόληση και το ΕΚΟΦΗΝ και την ισορροπία μεταξύ τους. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταφραστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου με μια αναπροσαρμογή της ρήτρα ε, ευελιξίας, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, δηλαδή το να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσει της λιτότητας σε έναν ε, κύκλο που δεν είναι τόσο ενάρρωτο όσο θα ήθελαν κάποιοι, αλλά που θα πρέπει να διορθωθεί που θα περιλαμβάνει και τους μηχανισμούς ευελιξίας που, με τους οποίους εξοπλιστήκαμε στο Six Pack, Two Pack και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο όλο αυτό το σύνολο νέων καινοτόμων εργαλείων που δεν έχουμε ακόμα αξιοποιήσει πλήρως όλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο για να το πω πιο σαφώς ε, ακούω στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία και αλλού ακούω να λένε αφού έχουμε λιτότητα και αυτή η λιτότητα φαίνεται να εδραιώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ίσως θα έπρεπε να ελευθερώσουμε λίγο τα επιτόκια ώστε να επανέλθουμε πιο αρμονικά, πιο ευέλικτα μέσα στον χρόνο. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ανοιχτεί αυτή η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και είναι σημαντικό, διότι πιστεύω ότι για να επιτύχει μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να βασίζεται σε έναν απλό διάλογο μεταξύ του εκάστοτε κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε σε καθολικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ως Ευρωζώνη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πρόβλημα έχουμε καθίσει σε μια κατάσταση λιτότητας από την οποία πρέπει να βγούμε. Τελευταία μου παρατήρηση, δεδομένου ότι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση στο γύρο τραπέζι σήμερα το πρωί που παρουσίασε ο κύριος Λαμασούρ, ανησυχούμε. Η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών δαπανών υπό τις τρέχουσες συνθήκες εφόσον μιλάμε για έναν προπολογισμό επενδυτικό και στον κοινωνικό τομέα, θα πρέπει να υποστηριχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εφόσον θέλουμε να μπούμε σε οδού, εξόδου από την κρίση, όχι ει βάρο της απασχόληση. Γι' αυτό το λόγο επιμένω είναι σημαντικό ειδικά για ορισμένα κράτη-μέλη, ειδικά για ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, αυτή η απέτηση δεν είναι τόσο προφανή. Αλλά εμεί, ε, στο πλαίσιο τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θεωρούμε ότι στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή θα πρέπει να δεσμεύσουμε κονδύλια υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Διότι γνωρίζουμε στι τοπικέ αρχέ, στι τοπικέ κοινότητε, αυτό που ονομάζουμε δαπάνε για υποδομέ είναι εξαιρετικά σημαντικέ ε, ε, προσφέρουν προβολή, ορατότητα, ε, δίνουν λόγο για την ύπαρξη του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Καταλαβαίνω στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή έχετε αρκετού αυτοκινητοδρόμου πια. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσετε και ορισμένου αυτοκινητοδρόμου πληροφοριών. Θα πρέπει να επενδύσετε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι εξίσου σημαντικό με τι υποδομέ. Αν όχι σημαντικότερο. Αυτό πιστεύω απορρέει από τις σημερινέ συζητήσει. Πραγματικά σας κάνω έκκληση να υποστηρίξετε αυτό το 25% που θα δεσμευτεί υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα το πω στον Επίτροπο Αντόρ ε, πόσο πολύ έχω υποστηρίξει αυτές τις, ε, αυτούς τους προσανατολισμούς. Σας ευχαριστώ ξανά όλες και όλους που παραστήκατε, που παραμείνατε στις εργασίες μας μέχρι το τέλος. Σας δίνω ραντεβού σε περίπου μισή ώρα, λίγο παραπάνω, στα σαλόνια, στους κατω, στον κατόροφο, για το δείπνο που θα σας προσφέρουμε εφόσον έχετε πρόσκληση, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι που βρίσκονται εδώ έχουν λάβει αυτό το περίφημο σας, για να παρευρεθούν στο δείπνο που θα προσφέρει ο Πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Μαρτίν Σούλτς, ε, όπου επίτιμος καλεσμένος ο επίτιμος ομιλητής θα είναι ο Πίτερ Πράτ, μέλος ε, του Προεδρείου της Κεντρικής Τράπεζας και που θα μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα στρατηγικών ανάπτυξης και δημιουργίας της συνεργασίας όπως υπό το πρίσμα μάλλον της Κεντρικής Τράπεζας. Σημαντικό ζήτημα. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι οι κονκάρδες που έχετε στη διαθέσή σας θα σας χρησιμεύσουν για να μπείτε στο κτίριο και για τη συνεδρίαση αύριο το πρωί. Λοιπόν, μην τις πετάξετε στα σκουπίδια, για, ώστε να μην χρειαστεί να ζητάτε άλλες αύριο το πρωί. Έχουμε ολοκληρώσει, ευχαριστώ ιδιαίτερο στους διερμηνείς και ραντεβού σε μισή ώρα. Γεια σας.